Okay, colleagues, please be Καθίστε αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε την απογευματινή μας συνεδρίαση. Έχουμε ενδιαφέροντα σημεία και στην απογευματινή ημερήσια διάταξη. Το πρώτο θέμα αφορά την εφαρμογή της κοινή διακήρυξης Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ της Βαρσοβίας. Θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τους ε, γνωστούς σε όλους μας καλεσμένους. Μάλιστα, με Ιδιαίτερα με τον Διευθυντή Κλόντ είχαμε συχνότατες επαφές, αλλά πρώτα θα δώσω το λόγο στον Διευθυντή Τίμο Κόστνερ για να μας μιλήσει για την αμυντική πολιτική. Είναι, Διευθυντής ε, Πολιτικής και Ικανοτήτων του ΝΑΤΟ και κατόπιν θα ακούσουμε τον κύριο Γκάμπορη Κλόντι που είναι στη Διεύθυνση Διαχείρισης Κρίσεων και Σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και το θέμα μας είναι γνωστό γιατί ήδη είχαμε την σχετική έκθεση εφαρμογής υλοποίησης και ε, τις 42 προτάσεις που υπευλήσαν από κοινού με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον κύριο Στόλτεμπεργκ και που αποτελούν τη βάση αυτή τη στρατηγική συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Θα δώσω το λόγο πρώτο στον ε, διευθυντή, τον κύριο Τίμο Κώστερ από τον ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να παραστώ στην Επιτροπή σας. Ε, πάντα είναι ευχάριστη η παρουσία μου εδώ και πάντα η παρουσία μαζί με τον Καμπουρή Κλόντι σε διάφορα περιβάλλοντα, όχι μόνο εδώ. Το θέμα μας ε, είναι η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κοινή δήλωση που υπεγράψαν πέρυσι οι τρεις και η οδός που ακολουθούμε για την υλοποίηση της κοινή δήλωσης. Η δήλωση υπεγραφή τον περασμένο Ιούλιο στη Βαρσοβία, όπως ξέρετε, και σε 6 Δεκεμβρίου πέρυσι, βάσει της κοινή δήλωσης, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και το ΝΑΤΟ και τα σχετικά συμβούλια ενέκριναν ε, ένα κοινό σύνολο 42 προτάσεων για την υλοποίηση της δήλωσης. Φυσικά η συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών είναι ουσιώδου σημασία στο σημερινό στρατηγικό περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ έχουν να αντιμετωπίσουν ε, προκλήσεις άνευ προηγουμένου και οι οργανισμοί μας έχουν ένα πλήρες σύνολο εργαλείων για να αντιμετωπίσουν μαζί τις προκλήσεις αυτές, κάτι που δεν μπορούσαν να κάνουν μόνες τους. Ε, θα ενισχύσουμε έτσι την ευρωπαϊκή άμυνα, κάτι που πρέπει να σημαίνει περισσότερα και καλύτερα μέσα των ευρωπαϊκών κρατών μελών, καλύτερη συνεργασία, περισσότερες αμυντικές δαπάνες, ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας και περισσότερη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας ε, αλλάζει το παιχνίδι στα, ε, της άμυνας ε, βελτιώνει τις ευρωπαϊκές δαπάνες, τις ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες και τα αμυντικά μέσα της Ευρώπης. Όλα αυτά είναι υπέρ του συμφέροντος της συμμαχίας. Ισχυρή ευρωπαϊκή άμυνα σημαίνει ισχυρότερο ΝΑΤΟ και πιο δίκαιο επιμερισμό των βαρών διατλαντικά. Και ισχυρότερο ΝΑΤΟ φυσικά σημαίνει και καλύτερη άμυνα της Ευρώπης. Καθώ επιδιώκει τι πρωτοβουλίε αυτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να ασφαλίσουμε οι προσπάθειε των δύο μερών να παραμείνουν συνεκτικέ και συμπληρωματικέ. Στη συνεργασία αυτή, το κοινό μα έργο, όπω έγινε το περασμένο χρόνο, έδωσε σημαντικά αποτελέσματα. Έχει αλλάξει ποιοτικά η συνεργασία μα. Ε, ε, η συνεργασία μεταξύ μα είναι πλέον κανόνα. Και μέσω αυτής ε, πιστεύω στέλνουμε ένα χειρό μήνυμα σε πολλούς αποδέκτες. Πρώτα απ' όλα προς τους δικούς μας λαούς και τους φορολογουμένους μας. Ότι δεν είμαστε ανταγωνιστικοί μεταξύ μας, ότι δεν σπαταλάμε τους ε, σπανίζοντες πόρους και ότι μεγιστοποιούμε την αξία μας μαζί. Και δεύτερον, ένα σημαντικό μήνυμα στους πιθανούς αντιπάλους μας, ότι παραμένουμε ενωμένοι, ώστε να μπορούμε να αντιδράσουμε στις προσπάθειές τους να αποδυναμώσουν τις κοινωνίες μας, διότι οι συνδυασμένες προσπάθειές μας φέρνουν ε, αποτελέσματα καλύτερα από ότι το άθροισμα των επιμέρους προσπαθειών μας. Και τέλος ένα μήνυμα προς εταίρους μας ότι πάντα είμαστε διατεθειμένοι να τους υποστηρίξουμε στην οικοδόμηση των δικών τους ικανοτήτων και μέσων και στη σταθεροποίηση της δικής τους γειτονίας που είναι και δική μας. Μέσα σε λίγους μήνες έχουμε επιτύχει απτά αποτελέσματα στην υλοποίηση των προτάσεων να επισημάνω κάποιες συγκεκριμένες δράσεις όπου πραγματικά σημειώθηκε πρόοδος. Πρώτα απ' όλα η συνεργασία για την αντιμετώπιση των ε, απειλών στον κυβερνοχώρο κάτι πολύ σημαντικό 10 από τις 42 ε, προτάσεις συγγνώμη τις υβριδικές απειλές 10 ε, προτάσεις λοιπόν σχετίζονται με την καταπολέμηση των υβριδικών απειλών. Η καλύτερη επίγνωση της κατάστασης είναι κρίσιμη σημασία για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απειλές αποτελεσματικά και η δημιουργία ε, ενός κέντρου αντιμετώπισης και ανάλυσης των υβριδικών απειλών ε, θα μας βοηθήσει ε, να έχουμε καλύτερη εικόνα της κατάστασης. Η συνεργασία με το εξή των στρατηγικών ομάδων θα μας βοηθήσει να στείλουμε ένα μήνυμα ότι παραμένουμε ενωμένοι υποστηρίζοντας κυρίως τους ανατολικούς μας εταίρους και στέλνοντας συντονισμένα μηνύματα και στα Δυτικά Βαλκάνια. Επίσης ε, θα συμμετέχουμε και θα συμβάλλουμε στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας για την καταπολέμηση των υβριδικών απειλών που συστάθηκε στο Ελσίνκι πρόσφατα. Δεύτερον, ε, συνεργασία και ο συντονισμός ε, επιχειρησιακά, κυρίως μεταξύ της επιχείρησης Σοφία και του Sea Guardian, ενισχύθηκαν με την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία στον τομέα της διοικητικής μέρημνας. Ε, αυτό βασίστηκε και στην παλιότερη εμπειρία στον Ινδικό ωκεανό όταν ασχοληθήκαμε με τις τρομοκρατικές απειλές εκεί. Οι πρόσφατες συντονισμένες κυβερναπειλές σε όλο τον κόσμο έδειξαν πόσο αδύναμες είναι οι κοινωνίες μας και τα θεσμικά μας όργανα και η συνεργασία, η εκπαίδευση, η άσκηση και η εκπαίδευση αναπτύσσονται ώστε να ενισχυθεί η συμπληρωματικότητα μεταξύ των διοργανισμών. Επιπλέον όσον αφορά τα αμυντικά μέσα, επιδιώκουμε να πετύχουμε συνοχή μεταξύ του σχεδιασμού στο ΝΑΤΟ και του σχεδίου ανάπτυξης δυνατοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συνεργασία μεταξύ των δύο ε, επιτελείων σε διάφορα επίπεδα της διαδικασίας αμυντικού σχεδιασμού συμβάλλει και η συμπληρωματικότητα των πολυεθνικών ε, προγραμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ επιδιώκονται με συγκεκριμένα αποτελέσματα, όπω για παράδειγμα στον τομέα του ενέργειου ανεφοδιασμού. Μετά, όσον αφορά την αμυντική βιομηχανία και έρευνα, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δημιουργήσει ένα μηχανισμό αλληλεπίδραση για περαιτέρω διάλογο σε βιομηχανικέ πτυχέ με εστίαση σε συγκεκριμένου τομεί κοινού ενδιαφέροντο. Για πρώτη φορά, το προσωπικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ από κοινού θα απαντήσουν σε ένα υβριδικό σενάριο στο πλαίσιο μια άσκηση οι προετοιμασίες όσον αφορά την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άσκηση CMX 17 τον Οκτώβριο, στην άσκηση αυτή του ΝΑΤΟ ε, και παράλληλα στην ΠΕΣ 17 έχουν προχωρήσει. Εκεί θα δοκιμαστεί η υλοποίηση η τρίτη, του ενός τρίτου των κοινών προτάσεων σε διάφορους δομικούς τομείς που έχουν εντοπιστεί από αφότερες πλευρές ε, όσον αφορά τη στρατηγική του ΝΑΤΟ και την συνεργασία προσωπικού σε θέματα όπως είναι η πρώιμη ε, ενημέρωση, η επίγνωση της κατάστασης, ε, η αντιμετώπιση των απειλών στον κυβερνοχώρο. Τέλος, ε, βοηθάμε τους εταίρους μας να ενισχύουν τα μέσα τους και την αντοχή τους, ειδικότερα στα Δυτικά Βαλκάνια και στην Ανατολική και Νότια γειτονία. Αυτό αποτελεί κοινό στόχο και των διοργανισμών. Η συνεργασία τόσο ε, στο πεδίο όσο και σε θέμα κεντρικών ε, επιτελείων ε, έχει πραγματοποιηθεί. Υπάρχουν επικοινωνίες στρατηγικές, αντιμετώπιση κυβερνητικών απειλών και η ασφάλεια σε κάποιες πιλωτικές χώρες όπως Βοσνία, Ζεγοβίνη, Μολδοβία, την Ισία. Λόγω της πολιτικής δέσμευσης ο διμερής διάλογος έχει επεκταθεί με διάφορες ε, υπουργικές διασκέψεις ε, υψηλού επίπεδου και προσκλήσεις σε αυτές με διάφορες ε, τυπικές και άτυπες συναντήσεις. Εγώ, για παράδειγμα, την περασμένη εβδομάδα παρευρέθη στη συνάντηση των Διευθυντών Πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ταλίν, στην Εστονία. Συμπερασματικά, να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι ούτε το ΝΑΤΟ ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν μόνοι τους. Κανεί μας δεν έχει μόνο του τα εργαλεία που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει τα θέματα ασφάλειας. Μαζί έχουμε ένα πλήρε σύνολο εργαλείων, το οποίο μπορεί να κάνει μια μεγάλη διαφορά. Και προσβλέπω στην περαιτέρω ανάπτυξη και ε, ένταση αυτή τη συνεργασία ε, ακόμη περισσότερο στο μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Θηδά. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον Διευθυντή της ΕΙΕΔ, τον κύριο Γκάμπορ Ικλόντι. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Χαίρομαι ιδιαίτερος ε, για την νέα ευκαιρία που έχουμε για ανταλλαγή απόψεων. Και χαίρομαι που είμαστε στο ίδιο με τον Τίμο. Όπως ε, είπε ο Τίμο, Προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε αυτό το σχέδιο. Δεν πρόκειται να επαναλάβω αυτά που είπα για την πορεία που ακολουθούμε. εγώ θα σταθώ σε μερικούς μόνο τομείς. Καταρχήν, τι γίνεται με την κοινή διακήρυξη της Παρσοβίας. Ήταν πολύ σημαντική αυτή η κοινή ε, διακήρυξη γιατί ε, αποτέλεσε το ορόσημο μιας αλλαγής της προσέγγισης ε, ε, που προκλήθηκε από τις γενικές αλλαγές στο ευρύτερο τοπίο. Και πυροδοτήθηκε αυτή η κοινή διακήρυξη μετά τη συνειδητοποίηση ότι αν θέλουμε ε, ουσιαστικές λύσεις και απαντήσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, ε, θα πρέπει αυτά τα δύο θεσμικά όργανα μετά από πολύ χρόνια δράνεια ως προς τη συνεργασία τους επιτέλους να συνεργαστούν και να συντονίσουν τις δραστηριότητές τους. Το 2014 πολύ συχνά το αποκαλούμε το έτος καμπή και αλλαγών μετά τις εξελίξεις ε, ανατολικά και νότια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το θέμα είναι ότι όχι μόνο οι ηγέτες μας, οι θεσμικοί ηγέτες ε, αναγνώρισαν ποιες είναι οι προτεραιότητες για τη δράση, αλλά αργότερα το Δεκέμβριο τα κράτη-μέλη αλλά και οι συμμαχοί μας ενέκριναν αυτές τις 42 προτάσεις, τη δέσμη των 42 προτάσεων. Και το θέμα δεν είναι μόνο αριθμητικά ότι τα 42 είναι περισσότερο από το 7 που ήταν αρχικά, άρα σημαίνει πρόοδο, Ε, βλέπουμε ποια κράτη-μέλη υποστηρίζουν αυτή την πρόταση. Δεν είναι μόνο η επιθυμία των ηγετών να συνεργαστούν αυτά τα δύο θεσμικά όργανα, αλλά ολόκληρη κοινότητα και το χωρονάτο και το χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στηρίζει αυτή τη συνεργασία. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι υπήρξε μία μετατόπιση της έμφασης σε ουσιαστική και πρακτική συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Όχι μόνο ε, στη θεωρία και στη, στον πολλαπλασιασμό των συνεδριάσεων και των συζητήσεων. Η, περιοχή, η προσοχή μεταστράφηκε σε πιο πρακτικά ρεαλιστικά βήματα και στην, ε, στην παρουσίαση έργου και αποτελεσμάτων. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι σημαντικό λοιπόν να δούμε τον κατάλογο των θεμάτων για τα οποία δόθηκε υπευλήθη έκθεση το προηγούμενο μήνα και στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Συμβούλιο του ΝΑΤΟ. Και μάλιστα ο κατάλογος αυτός είναι ενδεικτικός, δεν είναι εξαντλητικός. Δηλαδή δεν περιορίζεται μόνο σε 42 στοιχεία, 42 προτάσεις, κάνουμε τον έλεγχο και αν τα έχουμε υλοποιήσει τελείωσε και μείναμε ικανοποιημένοι. Είναι δεικτικό ο κατάλογος. Μερικές ιδέες μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω, να συμπληρωθούν από νέα στοιχεία, να διευρυνθεί ο κατάλογο των κοινών δραστηριοτήτων και ούτω καθεξής. Το Δεκέμβριο λοιπόν και όσο προετοιμαζόμαστε για το επόμενο ορόσημο που θα είναι το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου θα υποβληθεί η έκθεση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί κρατώντα αμύωτη την πίεση στα κράτη-μέλη, όχι μόνο στα θεσμικά όργανα, αλλά και στα κράτη-μέλη και στου συμμάχου μα, για να σκεφτούν, να στοχαστούν τι άλλο μπορεί να προσθεθεί και ποιε είναι οι συγκεκριμένε εξελίξει ε, που μπορούμε να αναφέρουμε. Όσο ετοιμαζόμαστε λοιπόν για το Δεκέμβριο, θα εκπονήσουμε την έκθεση για την περαιτέρω πρόοδο που έχει σημειωθεί και επίση θα γίνει συζήτηση ε, πώς μπορούμε να εμπλουτίσουμε αυτό το κατάλογο με νέα στοιχεία. Ένα σημαντικό τομέα θα είναι η αντιτρομοκρατία. Ε, ο πρόεδρος Τραμπ ήδη μίλησε ρητά για την ανάγκη του ΝΑΤΟ να επιδείξει έργο στην αντιτρομοκρατία. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι πολύ σημαντικό θέμα. Θα πρέπει λοιπόν να διαπιστώσουμε τι μπορούν να κάνουν από κοινού το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποφέρουν καρπούς. Και μάλιστα θα πρέπει να θεωρήσουμε αυτές τις δύο οργανώσεις όχι ως ξεχωριστές οντότητες, αλλά ως μηχανισμοί, ως εργαλεία στα χέρια των ενδιαφερομένων που είναι η κοινότητα των χωρών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει οι σύμμαχοι να διαπιστώσουν ότι υπάρχουν μηχανισμοί ώστε σε περίπτωση κρίσης αυτά τα διαθεσμικά όργανα να συνεργάζονται και να συντονίζονται. Σε ό,τι αφορά ένα άλλο θέμα που ανέφερε ο Τίμορ, τα μηνύματα. Το γεγονός ότι οι δύο οργανώσεις ε, ε, συνεργάζονται και μάλιστα προβάλλουν αυτή τη συνεργασία δίνει ένα πολύ ηχηρό μήνυμα προς το κοινό, τους εταίρους αλλά πιθανόν και τους αντιπάλους μας. Και μάλιστα αυτή η συνεργασία εξυπηρετεί και ένα στόχο αποτροπής και επίσης είναι και ένα μέσο για την πρόθεση της ανθεκτικότητας, γιατί δίνει το μήνυμα ότι η εργαλειοθήκη μας διευρύνεται. Έχουμε μια ολόκληρη κοινότητα που μένει συμπαγής ε, και συσπηρωμένη. Είναι σημαντικό λοιπόν να εμπεδώσουμε αυτό το μήνυμα και να το κρατήσουμε και για το μέλλον, ότι η κοινότητά μας είναι ενιαία και θέλει να παραμείνει ενωμένη. Σε ό,τι αφορά τα μέχρι τώρα αποτελέσματα. Ο τα ανέφερε ακροθυγός. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε συγκεκριμένους τομείς. Ένας είναι οι υβριδικές απειλές. Κατά τη γνώμη μας, ένα από τα μείζωνα αποτελέσματα ήταν η περσινή ίδρυση της μονάδας ανάλυσης υβριδικών απειλών, Hybrid Fusion Cell. Αυτή η μονάδα ανάλυσης συγκεντρώνει αποσπασματικές πληροφορίες, προειδοποιήσεις, ε, σήματα, από όλα τα θεσμικά όργανα, τα κράτη-μέλη και τους εταίρους μας, γιατί έχουμε ένα τεράστιο πλούτο πληροφοριών. Για παράδειγμα, μόνο τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ένα τεράστιο πλούτο ε, πληροφοριών. Η Γενική Διεύθυνση για την Ενέργεια, η Γενική Διεύθυνση Connect, ε, εσωτερικών υποθέσεων, έχουν ολόκληρες ε, αποθήκες πολύτιμων πληροφοριών. Οπότε η μονάδα ανάλυση υβριδικών απειλών ουσιαστικά συνδέει όλες αυτές τις αποσπασματικές πληροφορίες και όταν ε, εξετάζουμε συγκεκριμένα επεισόδια δεν βλέπουμε μόνο μία επίθεση στον κυβερνοχώρο ή μία προσπάθεια κινητοποίησης ε, του κοινού μιας χώρας για αντικυβερνητικές ε, διαδηλώσεις αλλά εμείς συνδέουμε τα κενά και διαπιστώνουμε αν υπάρχει ένα σχέδιο πίσω από όλα αυτά και αν όλα αυτά συνιστούν τμήμα μιας εκστρατείας γιατί τότε στοιχειοθετείται η έννοια τη υβριδικής απειλή. Οπότε αυτή η μονάδα ανάλυση βρυδικών απειλών συγκεντρώνει τι πληροφορίε, πραγματοποιεί την ανάλυση και δίνει την ευκαιρία στους ηθήνοντε ε, τη πολιτική να υποβάλουν συστάσεις είτε άμεσα προς την χώρα, την άμεσα ενδιαφερόμενη χώρα, είτε ε, ε διαπιστώνει χρειάζεται πανευρωπαϊκή αλληλεγγύη, επίδειξη αλληλεγγύη σε ένα θέμα, την ενέργεια αν είναι το θέμα αυτό. Επίσης, ε, δίνει ένα σημείο εισόδου-εξόδου προς το ΝΑΤΟ. Σε έναν ιδανικό κόσμο, και αυτό είναι το ζητούμενο, είναι να συστήσουμε μία κοινή εικόνα για τον εντοπισμό της κατάστασης. Δηλαδή, εμπειρογνώμονες και από το ΝΑΤΟ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μπορούν να ε, επεξεργάζονται τα ίδια στοιχεία και να διαμορφώνουν την ίδια εντύπωση. Αυτό είναι το απαραίτητο πρώτο βήμα. Μετά περνάμε στο δεύτερο βήμα, που αφορά την ε, εξακρίβωση του πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένη απειλή και μάλιστα με συγκεκριμένο τρόπο. Αυτά ως προς τη μονάδα ανάλυσης υβριδικών απειλών. Τώρα για να μην στα λέω και όλα ρόδινα, δεν είναι όλα καλά και άγια. Έχουμε ένα πρόβλημα. Αφορά την ε, ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών, εμπιστευτικών. Αυτό είναι ένα πρόσκομα και προσπαθούμε να βρούμε τρόπους να το παρακάμψουμε και να πραγματοποιήσουμε αυτή την ανταλλαγή και διαβαθμισμένων πληροφοριών, γιατί χωρί τέτοια ανταλλαγή δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεύτερο σημαντικό θέμα, πέραν των υβριδικών απειλών, είναι οι στρατηγικές, τα playbooks, τα εγχειρίδια στρατηγικής που μας λένε ε, σε ποιους κρίσιμους τομείς μπορούν να συνεργαστούν οι δύο οργανώσεις, ανταλλαγή πληροφοριών, ε, συγχρονισμός των τρόπων αντιμετώπισης κρίσης, ε, στρατηγική επικοινωνία. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Και μάλιστα αργότερα στο, στα πλαίσια του CMX και στα πλαίσια του PACE, που είναι οι παράλληλες και συντονισμένες ασκήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό θα κάνουμε, θα προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις ελλείψεις και τις αδυναμίες μας, όχι να τις ε, να θελοτυφλούμε, όχι να τις ε, παραχώνουμε και να κάνουμε όπως δεν τις βλέπουμε, αλλά να τις εντοπίζουμε και να τις διορθώνουμε. Και πάλι για τις ε, υβριδικές απειλές, ε, ιδρύσαμε και το Κέντρο Αριστείας για τις υβριδικές απειλές στο Ελσίνκι, που είναι και κάτι πρωτοφανέ. Είναι το πρώτο τέτοιο κέντρο αριστείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ευθύ εξ αρχή ε, το κέντρο αυτό είναι ανοιχτό και προ τα κράτη-μέλη και προς τους εταίρους μας από τον ΝΑΤΟ. Είναι το μοναδικό κέντρο αριστείας που λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ταυτόχρονα και για τις δύο κοινότητες, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ασχολείται με την έρευνα, τις ασκήσεις, την εκπαίδευση, ε, θέματα ασφάλεια τη θάλασσα, ασφάλεια τη ναυτιλίας. Το ανέφερε και ο Τίμορ. Εγώ θα επισημάνω δύο σημεία δεν μιλάμε μόνο για επιμελητιακή υποστήριξη και υποστήριξη μεταξύ των κεντρικών ε, υπηρεσιών, όπως υποσχεθήκαμε στη Βαρσοβία για την επιχείρηση Σοφία, κάτι που ήδη γίνεται και ήδη εφαρμόζεται. Υπάρχουν όμως δύο ενδιαφέρουσε εξελίξεις. Η μία αφορά ακριβώς την ανταλλαγή πληροφοριών. Και μάλιστα αφορά και τις κοινέ μας επιχειρήσεις και δραστηριότητες στο Αιγαίο κάτι που δείχνει και το πρόβλημα που έχουμε, δηλαδή την ε, δυσκολία ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών, αλλά επίσης διαπιστώνουμε ότι όταν υπάρχει θέληση βρίσκουμε και τον τρόπο να το κάνουμε. Ε, έχουμε επίσης ανάπτυξη εξωματοχών συνδέσμου και στα, στα, στα πλοία των επιχειρήσεων, ώστε μπορούν να δίνουν ε, εμπιστευτικές πληροφορίες και να λέει, κοιτάξτε εκεί, 200 μίλια από εδώ, είναι ένα πλοίο που καλό θα ήταν να το ελέγξουμε ή μέσω των ε, πρωτευουσών. Είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Αν υπάρχει επιθυμία και βούληση, θα βρούμε τρόπο για την ανταλλαγή των πληροφοριών. Τζέφρι, άφησε τον καλεσμένο μας να ολοκληρώσει, παρακαλώ. Και ακόμη πιο ενδιαφέρον και σημαντικό στο μέλλον είναι το γεγονός ότι Έχουμε δύο οργανώσεις που ουσιαστικά ενεργοποιούνται στον ίδιο τομέα και οι δύο οργανώσεις αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα της έλλειψης πόρων, το, πολύ, το, το κόστος ε, της διατήρησης ε, των στοιχείων τους και το κόστος του απόλυτου διαχωρισμού των δραστηριοτήτων των ε, δύο οργανώσεων είναι ακόμη πιο μεγάλο. Οπότε μπορούμε ίσως με πιο ελαστικό τρόπο να αξιοποιούμε από κοινού τους πόρου, κάτι που ήδη συμβαίνει σε μερικές περιπτώσεις. Και μάλιστα έτσι με τέτοια συνεργασία νομίζω θα εξυπηρετούμε καλύτερα και τους εταίρους μας, τους άμεσα ενδιαφερομένους. Αυτά για τη θάλασσα, για την ασφάλεια στη θάλασσα. Και τέλος, για τη δημιουργία ικανοτήτων. Ο μίλησε για τα τρία πιλωτικά προγράμματα, τις τρεις πιλωτικές υποθέσεις. Προσπαθούμε να βρούμε πώς θα αποφύγουμε τη σύγκρουση αρμοδιοτήτων και να δημιουργήσουμε συμπληρωματικότητα. Γιατί μόνο επί τόπου πηγαίνουμε και βλέπουμε «Α, είμαστε και οι δύο παρόντες για το ίδιο πράγμα». Υπάρχει επικάλυψη. Θα πρέπει λοιπόν να συντονίζουμε και τα σχέδιά μας και εκ των προτέρων, όχι μόνο σε τελευταία φάση εφαρμογής. Έτσι θα είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί. Γι' αυτό και έχουμε τι τρει πιλωτικέ υποθέσει με διεύρυνση του πεδίου των χωρών και των σχεδίων. Και θα συνεχίσουμε με βάση την εμπειρία που θα αποκομίζουμε. Επίση, στο πλαίσιο των υπηρετικών απειλών προσπαθούμε να βοηθήσουμε τι χώρε εταίρου να αναπτύξουν την αθεκτικότητά του. Ξεκινήσαμε με τη Μολδαβία. Μόλι ολοκληρώσαμε την σχετική έκθεση και την επόμενη, εβδομάδα. Ε, την επόμενη Δευτέρα θα πάμε στην ε, Γεωργία για τη δεύτερη έκθεση και ίσως το φθινόπωρο στην Ιορδανία. Και στις τρεις χώρες ε, είναι παρόν και το ΝΑΤΟ και ήδη είχε σημαντικές δραστηριότητες. Οπότε έχουμε και άλλες ευκαιρίες να συσπυρώσουμε, τις, να συνενώσουμε τις δυνάμεις μας. Και μερικές φορές όταν είμαστε παρόντες στις ε, χώρες εταίρους ε, με έντονο τρόπο, είμαστε πιο ορατοί, τα αποτελέσματα είναι καλύτερα, άλλες φορές είναι καλύτερο να είμαστε πιο διακριτικοί και παρασκηνιακά να συντονίζουμε τις προσπάθειές μας ώστε να εξασφαλίζουμε την συμπληρωματικότητα. Άλλε φορές η προβολή βοηθάει και άλλε όχι. Και όπως σας είπα, ε, μέχρι το Δεκέμβριο θα αναπτύξουμε και άλλες ιδέες, κυρίως σε δύο τομείς. Ο ένας αφορά την αντιτρομοκρατία και ο δεύτερος την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Και στους δύο τομείς, με βάση και την καθημερινή μας πείρα, ξέρουμε ότι χρειάζονται πρακτικές λύσεις και για τους δύο Βέβαια, ωραία και εύκολα τα λόγια, τα έργα είναι πιο δύσκολα. Έχουμε περιορισμού ό,τι αφορά την καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Το πρώτο είναι η ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών. Εκεί έχουμε πρόβλημα. Είναι εμπιστευτικέ οι πληροφορίε. Επίση, δημιουργία ικανοτήτων σε τρίτε χώρε. Θα μπορούσε να μα βοηθήσει στην καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Στον κυβερνοχώρο έχουμε πολλά πράγματα, πολλέ δυνατότητε, κοινέ ε, ασκήσει, κοινά συστήματα εκπαίδευση η κατάρτιση, επίσης ε, θέσπιση συγκριτικών κανόνων ή για τις κοινέ αποστολές και επιχειρήσεις. Μερικές φορές ε, οι χώρες, ανάλογα με το που αναπτύσσουν τις δυνάμεις τους, ακολουθούν διαφορετικά πρότυπα. Πάντως, ε, σε αυτούς τους δύο τομείς θα έχουμε εύκολα πρόοδο, σχετικά εύκολα, απλώς θα πρέπει να μεριμνήσουμε, να κρατήσουμε αυτή την όθηση που έχουμε πάρει τη φόρα που έχουμε πάρει σταθερή και να επεξεργαζόμαστε, να ασχολούμαστε κυρίως με απτά και ρεαλιστικά σχέδια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. για την εισαγωγή αυτής της συζήτησης που μας προσφέρετε. Και φυσικά αυτό σχετίζεται και με την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ε, Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ. Η κυρία Καηλή, πρόεδρος της ΔΥΝΑ, την εδώ παρούσα. Θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ για την ε, πρόληψη αυτής της πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δεν είμαι εδώ από την αρχή, αλλά θέλω και εκ μέρου τη ε, κοινοβουλευτική ε, αντιπροσωπεία στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να σα ε, καλωσορίσω και εγώ και να σα ευχαριστήσω. Θα ήθελα να διατυπώσω κάποιε ερωτήσει, αλλά φαντάζομαι ότι δεν μπορείτε να ξεπεράσετε τα όσα είπατε και να μα δώσετε πιο πολλέ πληροφορίε. Θα προσπαθήσω πάντω. Η συνεργασία Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ είναι για μα ένα από του πυλώνε μια ενεξελίξη πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την ασφάλεια και την άμυνα και δεν πρέπει να σταματήσουμε αυτές τις ομιλίες αλλά να τις συνεχίσουμε για να προσπαθήσουμε να διαγνώσουμε το πεδίο συνεργασίας που απλώνεται μπροστά μας γιατί έχουμε και θέματα άμυνας ασφαλών. Καλώς ορίζω φυσικά την έκθεση εφαρμογής ε, από πλευράς των δύο ε, οργανισμών που δημοσιεύτηκε πριν από δύο εβδομάδες ε, και θα ήθελα να διατυπώσω κάποια σχόλια για την υλοποίηση υπογραμμίζεται στην έκθεση ότι η λογική, δυναμική, ποιότητα ε, των ε, τη συμμετοχή μα, τη προσήλωσή μα σε αυτή τη συνεργασία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και ο κύριος Στόλτενμπεργκ επίση την υπογράμμισε, ιδιαίτερα στην επίσκεψη το Μάιο. Θέλετε όμως παρακαλώ, να μου δώσετε περισσότερε λεπτομέρειες, αλλαγή νοοτροπίας λέτε, ποιότητα, δυναμική, δηλαδή θέλουμε κάτι πιο συγκεκριμένο εδώ. Αυτό θέλετε να μας πείτε. Και επίσης, αναφέρατε και εσείς ξεκάθαρα ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης της, διοργανικής, της ε, συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών ε, ως προς την ανταλλαγή πληροφοριών. Ε, θέλετε να μας δώσετε πιο πολλές πληροφορίες σε σχέση με την αξιολόγηση μιας ε, σχεδιαζόμενης ε, ανταλλαγής πληροφοριών και πώς με αυτή μπορεί να βελτιωθεί η καταπολέμηση των ευρυδικών απειλών, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν χώρες που δεν είναι διτεθειμένες να προβούν σε αυτή την ανταλλαγή απόψε, να έχετε βρει κάποιο πεδίο συνεννόησης με βάση το οποίο μπορεί να υπάρξει αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών. Ε, θέλετε βοήθεια, μπορούμε εμεί με τι συζητήσει μα εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσουμε και επίση για τη θαλάσσια ασφάλεια και τη, Μεσόγειο έχουμε για την παγκόσμια θαλάσσια ε, ασφάλεια, ασφάλεια θαλάσσιες μεταφορές, αποφασίσει να, να πραγματοποιήσουμε συμπληρωματικές δράσεις από την εμπειρία σας με το Frontex, το Τρίτον, το Σοφία αλλά και τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ. Όλη αυτή η συνεργασία βλέπετε να φέρνει ήδη ε, την υλοποίηση κάποιων συγκεκριμένων στόχων, ε, κοινών στόχων βεβαίω. και ε, πιστεύετε ότι μπορούμε να την ενισχύσουμε αυτήν την υλοποίηση των κοινών στόχων. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Φαντάζομαι ότι και η Αν Γκόμε, μόλις σταματήσει να βγει θα μπορέσει να σα κάνει μια πολύ επίκαιρη και σημαντική ερώτηση. Ε, εν τω μεταξύ ο κύριο Γκάλερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ τους δύο μιλητές. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω εδώ. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η συνεργασία. Φυσικά και εγώ πάντα υπεστήριζα αυτή τη συνεργασία με τις 42 προτάσεις. Ως πολιτικός θα ήθελα κάποια στιγμή να μπορώ να πω α, ένα, δύο, τρία τα έκανα, τα κατάφερα, υλοποιηθήκανε. Και έτσι μπορώ να πω και στο ψηφοφόρο μου, να, αυτό το υποστήριξα και το καταφέραμε και όλα να το επιτύχουμε. Ξέρω ότι μπορεί να είναι ίσως πρόωρο να σας ζητάω κάτι τέτοιο. Αλλά υπάρχει κάποια σχετική πρόθεση, δηλαδή να κοιτάτε ένα τα θέματα και να βλέπετε ή να επιβλέπετε την υλοποίησή τους. Και βέβαια προτεραιότητες. Αυτά τα 42 σημεία προχωρούν εκ παραλίλου όλα. Υπάρχουν προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΝΑΤΟ προς τη μία την άλλη Και για τον κύριο Ινκλουντή δεν ξέρω εάν θα συμφωνήσω στον τρόπο με τον οποίο περιγράφεται τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των δύο παράλληλων ε, αυτών αποστολών στο ίδιο πεδίο. Εγώ θα προτιμούσω είτε πρόκειται για τον ε, κόλπο της Γουινέας, είτε πρόκειται για την Μεσόγειο και ιδιαίτερα αφού οι Αμερικανοί δεν ενδιαφέρονται και δεν εμπλέκονται σε δραστηριότητες στον τομέα αυτών. Εγώ λοιπόν θα προτιμούσα να λαμβάνουμε την απόφαση ποιος εκ των δύο αναλαμβάνει τη δράση. Δεν χρειάζεται να είναι και οι δύο παρόντες, ο, επιπλέον αναγκαίος συντονισμός. Πριν αρχίσουμε λοιπόν, να αποφασίσουμε ποιος το αναλαμβάνει. Και θα έχει υποστηρικτική δράση, επικουρική δράση ο άλλος, δορυφορικές εικόνες φέρει είναι κάτι άλλο που μπορεί να προσφέρει. Αλλά ο ένας από τους δύο, όχι και οι δύο ταυτόχρονα στο ίδιο, πεδίο δράσης. Και μια τελευταία ερώτηση Αντίθετα από τον ΝΑΤΟ, εμεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε και νομοθετικέ αρμοδιότητε. Επομένω, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατυπώνει προτάσει, οδηγούν αυτέ σε νομοθεσίε, σε τομεί που έχουν να κάνουν και με την πιστοποίηση, την τυποποίηση, τι τεχνικέ προδιαγραφέ ή πρότυπα. Έχουμε προχωρήσει αρκετά στη συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Μάλλον όχι, μάλλον όχι αρκετά. 60 χρόνια τώρα έχουμε συνεργασία, αλλά δεν έχουμε μπορέσει να εξασφαλίσουμε αυτή τη διαλειτουργικότητα των προτύπων και των πιστοποιήσεων μα. Εάν λοιπόν το θέμα είναι η πιστοποίηση, α διατυπωθούν συγκεκριμένε ε, νομοθετικέ προτάσει για να ε, καταργηθεί αυτή η προπόθεση ένα συγκεκριμένο κομμάτι στρατιωτικού υλικού, όπλου, εργαλείου κτλ. να χρειάζεται πιστοποίηση μετά την πρώτη ε, πιστοποίηση σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό πρέπει να υπάρχει ως δεδομένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την πολιτική προστασία ένα ε, εργαλείο ή ένα όπλο που έχει παραχθεί στο Ρωμένο Βασίλειο να γνωρίζεται ως πιστοποιημένο και σε όποια άλλη. Αλλά στο στρατιωτικό τομέα δεν το έχουμε αυτή την αμοιβαία αναγνώριση. Εάν λοιπόν παράγεται κάτι και πιστοποιείται σε μια χώρα και μετά πρέπει να εξαχθεί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από ό,τι μου λένε δηλαδή, θα πρέπει να περάσει από τη διαδικασία της αναγνώρισης και πιστοποίησης και σε κάθε άλλη χώρα στην οποία θα πρέπει να μπει. Ας κάνουμε λοιπόν κάτι νομοθετικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και διευκολύνουμε έτσι και τον ΝΑΤΟ αφού δεν έχει αυτό ε, νομοθετικές εξουσίες. Ευχαριστώ, λέει και η Πρόεδρος. Κυρία Γκόμες, μπορεί τώρα να μιλήσει, να περιμένουμε λίγο ακόμα, να πάρετε μια ανάσα. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για τις ε, ε παρουσιάσεις, εξηγήσει και εγώ καλωσορίζω την ε, πρόταση, με, την ε, δήλωση με τις, 52, με τις 42 προτάσεις σημειώνουμε πρόοδο πρέπει να πω χάρη σε αυτήν. Μπορούμε έτσι περαιτέρω να προχωρήσουμε και στους τομείς όπου έχουμε ασφαλώς ε, μεγαλύτερη συνεργασία ή διαδραστική σχέση και μπορούμε και αυτή να την ενισχύσουμε. Ε, θα έλεγα πριν κάνα δύο χρόνια ότι για το Κυπριακό το Κυπριακό αποτελούσε πρόσκομα στην συνεργασία τώρα και ότι δεν έχει ακόμα επιληθεί το Κυπριακό, αν και κάνω, διατυπώνω κάθε ευχή ώστε να ευοδοθούν οι προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα των Εθνών για την εξέβρεση λύσης. Τώρα όμως έχουμε μπορέσει να προχωρήσουμε. Μπορείτε λοιπόν να μας ενημερώσετε πώς έγινε αυτό. Ξέρω μένω ότι στην πράξη υπήρχαν αλλαγές προς το καλύτερο. Αλλά τώρα έχουμε περάσει ένα άλλο επίπεδο συνεργασίας και διάρθρωσης. Επίσης, Μας είπατε τα, κάτι το αρκετά συγκλονιστικό. Δεν ε, είχα την εντύπωση τόσο ότι από τόσο μα είπατε λέει, το πρόβλημα οφείλεται στη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, αλλά με, από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση προέρχονται τα προβλήματα. Αναφερθήκατε σε τόσε διαφορετικέ και αλληλοσυγκρουόμενε ή αποκομμένε μεταξύ του πληροφορίε και ε, συμπεριφορέ από διάφορε γενικέ διευθύνσει Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι πραγματικά συνταρακτικό. Ε, και πολύ εντυπωσιακό ω πληροφορία. Μπορεί αυτό να οδηγήσει με την αναγνώριση και εντοπισμό των προβλημάτων σε αντιμετώπιση, σε πιο συντονισμένη δράση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ένα άλλο. Πώς πραγματοποιεί τη στρατηγική επικοινωνία σε συγκεκριμένε ε, υποθέσεις. Η Πορτογαλία, πατρίδα μου, πριν από δύο εβδομάδες, την προηγούμενη ακόμα, γνώρισε τραγικές σκηνές με μια τεράστια επίθεση εναντίον ενός, μιας αποθήκης εξοπλισμών οπλικών, οπλισμών της Πορτογαλίας και μάλιστα πολύ σημαντική και για τον ΝΑΤΟ αλλά και για την παγκόσμια ε, ασφάλεια. Πώς θα αντιμετωπίσετε λοιπόν κάτι τέτοιο και ξέρω ότι δεν αφορά ένα κρατός μέλος μεμονωμένο αλλά και άλλα κράτη-μέλη έχουν γνωρίσει, ακόμα και επιθέσει σε στρατιωτικές βάσεις τους. Και μάλιστα οι αμερικανικέ βάσει υπό τον έλεγχο των Αμερικανών, ε, Γερμανία, Φιλιππίν. Η επικοινωνιακή κάλυψη μια τέτοια ε, περιστατικού Πώ καλύπτεται. Πόσο εξασφαλίζεται. Επίσης αναφερθήκατε στη σημασία της στρατηγικής επικοινωνίας με τη Δυτική Βαλκανική. Και εδώ θέλω κάποιες πληροφορίες συγκεκριμένε, γιατί ακούω αρκετά ανησυχητικά ενισχυτικές ειδήσει ως προς την ανάδειξη των λεγόμενων μουτζαέντιν του λαού στην Αλβανία. Αυτοί οι μουτζαέντιν που ξέραμε ότι αναπτύσσουν τις δραστηριότητε τους στο Ιράκ με, με βλέψεις συγκεκριμένα στο Ιράν, προχωρούν από το Καμχούρια, περνάνε στην Αλβανία και φαίνεται να Ξενών αρκετές δυσκολίες, ταραχές, προβλήματα με χρηματοδότηση βεβαίως Σαουδικής Αραβίας και μπορούμε να υποθέσουμε και διαφόρων άλλων. Ε, όχι, αν μπορείτε, αν λοιπόν ε, να μας ενημερώσετε αν αυτή η επικοινωνιακή διαχείριση φέρνει τους απαιτούμενους καρπούς και αν είναι αίσθητο, θα ήθελα να ξέρω, για την Τουρκία και το Αιγαίο. όπου βλέπετε ότι υπάρχουν σημαντικές, ε, σημαντικά ωφέλη από τις επιχειρήσεις στο Αιγαίο. Δεν το συζητεί κανείς, αλλά υπάρχει μια σταθερή ροή περί των 100 ανθρώπων την ημέρα. Αυτοί τώρα μετανάστες τους πούμε, πρόσφυγες τους πούμε, δεν θεωρώ ότι είναι απειλή, δεν συνιστούν απειλή, ευκαιρία μόνο και με αυτή την ροή. Μια ροή λοιπόν 100 την ημέρα. Σταθερή ροή. Κανείς δεν την αναφέρει. Όλοι μιλούν ε, για τη σκοτεινή αυτή συμφωνία με την ε, Τουρκία ότι φέρει αποτελέσματα. Αλλά δεν έχει φέρει κανένα αποτέλεσμα. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε εσείς μέσα από τη διάρθρωση του ΝΑΤΟ πώς αντιλαμβάνεστε αυτή την κατάσταση. Τζέφρι Ευχαριστώ πρόεδρε. ευχαριστώ τους δύο μιλητές μας. Βεβαίω θα πρέπει να σας επισημάνω, όχι βέβαια για τη δική μας την Επιτροπή, αλλά γενικά για το Κοινοβούλιο, ότι υπάρχει εντύπωση στους ορισμένους βουλευτές ότι αν δεν κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν το κάνει κανείς άλλος. Δηλαδή ότι θα προκύψει κενό ασφάλειας και άμυνας, το οποίο μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να καλύψει. Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι κανείς δεν πράττει τίποτα σε αυτό. Ότι ξεκινάμε από το μηδέν. Με αυτό το πράγμα που ονομάζεται ε. ε. Εγώ πιστεύω ότι συνιστά και απόλυτη πόρων η εμπλοκή σε διάφορε δραστηριότητε τη ΕΕ. Υπάρχουν κράτη, πλην τη Κύπρου βεβαίω και τη Μάλτα, όλα τα κράτη είναι στο τραπέζι του ΝΑΤΟ με κάποια ιδιότητα. Ε, ή τέλο πάντων έχουν κάτσει στο τραπέζι του ΝΑΤΟ, έχουν συμβάλει σε επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, πλην της Κύπρου και της Μάλτας. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει πόρους ή στρατιωτικές δυνατότητες που να μην έχει το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, βλέπω να έχουμε μπει σε μια νέα ε, οργουελική φάση ρητορίας που πια γίνεται πιστευτή γιατί από όλου ή από του περισσότερου, γιατί επαναλαμβάνεται τόσο συχνά που την πιστεύουμε, την ακούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπρόσωπο, ένα ο άλλο, μπράβο καλά τα κάνατε, επένου ανταλλάσσουν και Τελικά τα πιστεύει και ο κόσμο. Πολύ επικίνδυνο, πολύ επικίνδυνο. Και θα ήθελα να δείτε πόσο δύο ερωτήσει. Για την κυβερνό, κυβερνό απειλή. είναι ο συγκεκριμένο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τι μπορεί να συμβάλλει ναυτικές επιχειρήσεις στη Μεσόγειο. Υπάρχει κάποιος, ε, κάποια, ηγετική, διοικητική αρχή διοικητής στις ναυτικές αυτές επιχειρήσεις που να μπορεί να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις. Βλέπω και διαφωνώ απολύτως με την ε, συνάδελφο κυρία Γκόμες ότι δεν υπάρχει καμία οργάνωση. Έχουμε δηλαδή καταλήξει σε μια λύση καταστροφική, η οποία θα οδηγήσει ακόμα, σε ακόμα χειρότερα αποτελέσματα. Και βλέπουμε ότι όλο και, περνούν, όλο και περισσότεροι περνούν τη Μεσόγειο, διασχίζουν τη Μεσόγειο. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν αντιδρούμε, γιατί, δεν, γιατί περιμένουμε να μπουν στα πλοιάρια αυτά με στο νερό οι άνθρωποι αυτοί για να αντιδράσουμε, γιατί να μην τους δίνουμε εισιτήρια από τις χώρες της Βόρειας Αφρικής να έρχονται με ασφάλεια αεροπορικός. Μας λένε ότι, μας είπαν το πρωί ότι είναι 500.000 αυτοί που βρίσκονται στη Λιβύη και περιμένουν να μπουν σε πλοιάρια και άλλοι πολλοί που έχουν πάρει ήδη το δρόμο. Σε κάνα δύο χρόνια δηλαδή όταν καταστεί ανυπόφορη πια η καταστροφή, θα ξυπνήσει ο κόσμος. Αλλά θα είναι αργά. Πρέπει να σταματήσουμε, πρέπει να κλείσουμε την πόρτα και να πούμε δεν δεχόμαστε άλλους παράτυπους μετανάστες σε χώρες ευρωπαϊκές, τελεία και παύλα, γιατί αν δεν το πει ή όσο δεν το έχει πει αυτό κανείς, ό,τι νόμους και συμβάσεις, γιατί πρέπει να αλλάξει και αυτό βεβαίως για να μην αντιμετωπίζουμε διαρκείς ε, ε, δικαστικούς αγώνες από τους κρατικοδίαιτους δικηγόρους μας. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουν και οι συμβάσει διεθνεί κλπ. Αλλά θα βρεθούμε από μια καταστροφή αν δεν αλλάξουμε. Και πρέπει και αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι αναλαμβάνουν τις επιχειρήσεις ε, στο ναυτικό πεδίο να είναι πεπισμένοι για το όφελο και τη χρησιμότητα των επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν. Επίσης, ε, η αμυντική σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου, ως τελευταία ερώτηση, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς πιστεύετε ότι θα διαμορφωθεί. Και ευχαριστώ πολύ. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν ε, ιδανική η κατάσταση, τουλάχιστον όπως βλέπω εγώ τα πράγματα, λέει η Πρόεδρος. Θα ήθελα να, ακούσω σχόλια. από τους ομιλητές μας, αν και ξέρω ότι είναι δύσκολο ε, για κάποιον που δεν ε, υπάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει με τον ίδιο τρόπο δηλώσεις ή σχόλια. Αλλά το Κοινοβούλιο αυτό είναι, οι διαδικασίες του αυτές είναι. Εμείς αποφασίζουμε Υπάρχουν διαδικασίες που ακόμη δεν έχουν εκριθεί. Έχει αποφασίσει ένα πρώτο δηλό βήμα του Συμβουλίου για ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας που συμβάλλει στην ανάπτυξη, που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των κοινών μας προσπαθειών για την κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα και οι πρώτες νομοθετικές απόπειρες που ξεκινούν με μια καταχώρηση σε, Μητρό και που είδαμε ύστερα από πολλές προσπάθειες της ΕΝΤΕ να προχωρήσει στην Μήτρε μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως θα πρέπει να επαγρυπνούμε ώστε να μην επαναλαμβάνεται η δουλειά, να μην έχουμε επικαλύψεις δηλαδή, οι ασυμβατότητες, αλλά ό,τι δουλειά γίνεται να γίνεται κατά τρόπο συμπληρωματικό. Η προσέγγιση όπου από την απόψη της ασφάλειας είναι τελείως διαφορετική από αυτήν της προσέγγισης που στόχο έχει την ενίσχυση της βιομηχανίας και θα πρέπει και αυτό να το λάβουμε υπόψη. Και να βρούμε και τις αυτονόμιες δυναμικές και τις προσπάθειες για να επισκοπήσουμε τις δυνατότητες και μόνο κάποιες σκέψεις ήταν αυτές ύστερα από τις χτεσινές τις σημερινές πρωινές και μεσημεριανό απογευματινές συνομιλίες στα θέματα αυτά Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί λοιπόν και να βρούμε αυτή την, ε, αυτό το πνεύμα συνεργασίας, γιατί είναι ένα θέμα λεπτό, ένα θέμα σοβαρό, ένα θέμα σημαντικό και απαιτεί μεγάλο βαθμό υπευθυνότητας και ιδιαίτερο και από το Κοινοβουλίο. Έχετε το λόγο. Έχετε το λόγο. Δεν ξέρω ποιον κύριο εννοείται ακριβώς, γιατί είμαστε και πολλοί. Ευχαριστούμε για όλα τα σχόλια και όλες τις ερωτήσεις σας. Ε, ε, κάποια πράγματα τα πεθαίνετε στον Γκάμπορ, αλλά θα απαντήσω και εγώ σε κάποια πράγματα που θεωρώ σημαντικά από αυτά. Πρώτα απ' όλα, η φιλοσοφία και η ποιότητα της συνεργασίας μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ανταλλαγή πληροφοριών και κάποιες από τις δυσκολίες ε, που σχετίζονται με όλα αυτά. Όταν λέμε αλλαγή νοοτροπίας, δεν μιλάμε απλά για μια συμφωνία ανταλλαγής πληροφοριών. Από πολλές απόψεις ε, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Ε, αυτό σκεφτόμαστε όταν προκύπτει οτιδήποτε λέμε μπορούμε, ε, εξορισμού να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση αντί να προσπαθήσουμε πρώτα απ' όλα μόνοι μας και μετά να σκεφτούμε α, μήπως ε, ε, να δούμε τι κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε υπάρχει μια συνεχής σχεδόν αυτόματη τέτοια αντίδραση ότι πριν αρχίσω να σχεδιάζω οτιδήποτε, οποιαδήποτε λύση για οτιδήποτε σήκωνω το ακουστικό και παίρνω τον κάμπορ ή οποιονδήποτε άλλο συνάδελφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπω τι κάνει η άλλη πλευρά, τι μπορούμε να συνδυάσουμε ε, πόσα είναι δυνατόν να κάνουμε μαζί δεδομένων των θεσμικών περιορισμών που έχουμε. Αυτά όσον αφορά την οτροπία. Όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, να εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίε. Αλλά η κυρία Γκόμε ε, ε, ρώτησε πώ είναι δυνατόν να επιτεθεί τόση πρόοδο. Για να είμαι ειλικρινή, το μεγαλύτερο μέρο τη συνεργασία γίνεται μεταξύ μελών του προσωπικού. Όσο λοιπόν δεν είμαστε σε επίπεδο συμβουλίου προ συμβούλιο ή κράτο προ κράτο, αποφεύγουμε τις θεσμικές δυσκολίες. Μεταξύ μελών του προσωπικού δεν έχουμε και πολλούς περιορισμούς. Συζητάμε άνετα μεταξύ μας. Εντάξει υπάρχουν κάποια επίπεδα διαβάθμισης ε, όπου δεν μπορούμε να μοιραστούμε πληροφορία μεταξύ μας. Αυτό είναι και μονόδρομο το πρόβλημα γιατί στο ΝΑΤΟ διαβαθμίζουμε περισσότερες πληροφορίες και σε υψηλότερη διαβάθμιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά αντίστοιχα έγγραφα, για παράδειγμα το έγγραφο υλοποίηση των 42 προτάσεων, είναι το ίδιο έγγραφο και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δημόσιο, σε μας είναι περιορισμένο. Οπότε δεν τα έχουμε λύσει όλα και ούτε οι καταστάσει όλε είναι ιδανικέ, αλλά η πρόοδο που έχει σημειωθεί ε, έχει επιτευχθεί κυρίω σε επίπεδο προσωπικού. Τώρα, σε έναν ιδανικό κόσμο, το καλύτερο θα ήταν να κάνουμε και μεγαλύτερη πρόοδο μεταξύ κρατών, μεταξύ συμβουλίων. Αυτό είναι προβληματικό, αυτό είναι δύσκολο, διότι έχουμε αυτού τους θεσμικού ε, περιορισμούς που μας το απαγορεύουν και εδώ δυστυχώ δεν είναι κάτι στο οποίο μπορώ να δώσω λύση εγώ. Οι κυβερνήσει, τα κράτη πρέπει να το λύσουν μεταξύ του. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό ότι πάντα υπάρχουν τρόποι να παρακάμψουμε τα εμπόδια. Κάτι που προωθούμε, για παράδειγμα, Συζητώντα με τα διάφορα κράτη, τους λέμε μην περιμένετε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ να ανταλλάξουν διαβαθμισμένε πληροφορίε μεταξύ τους. Αν εσείς ω κράτος διαθέσετε και στους δύο ταυτόχρονα αυτές τις πληροφορίε, δεν χρειάζεται να γίνει ανταλλαγή μεταξύ μας. Οπότε εκεί, χωρί να αλλάξει καμία διαβάθμιση, ούτε καμία νομοθεσία, μπορείτε να διευκολύνετε τι ζωέ και των διοργανισμών. Ε, γίνεται δηλαδή μια ε, αξιοσημείωτη προσπάθεια. Τώρα η ερώτηση του κ. Γκάλερ, η υλοποίηση πότε γίνεται και ποια είναι οι προτεραιότητε. Θα έχετε δει την έκθεση υλοποίηση, φαντάζομαι, θα έχετε δει τι τρέχει αυτή τη στιγμή, απομένουν πολλά να γίνουν. Δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε κάποιο σημείο που θα πούμε ορίστε εδώ τελειώσαμε. Διότι ο στόχο που έχουμε μπροστά μα είναι κινούμενο όλο και περισσότερα ζητήματα ανακύπτουν, όλο και περισσότερα θέματα στα οποία μπορούμε να συνεργαστούμε. Για παράδειγμα, η πρόοδος που σημειώνει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ευρωπαϊκή Αμυντική Συνεργασία ε, μας δείχνει ότι υπάρχουν πολλοί νέοι τομείς όπου μπορούμε να συνεργαστούμε. Προσπαθούμε λοιπόν εμείς να ε, λαμβάνουμε υπόψη όσο γίνεται περισσότερα ε, σημεία αυτή της λίστας, ε, αλλά είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και άλλα. Και αυτό με φέρνει ε, στην ερώτηση του κ. Βανόρντεν, που αφορά την ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική και τους πόρους που δεν ανήκουν μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή μόνο στα κράτη-μέλη. Να πω ότι το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο και η ΠΕΣΚΟ αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. ότι δημιουργούν ε, νέες δυνατότητες, νέα μέσα, νέους οικονομικούς πόρους ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι χρήματα που βγαίνουν από τον αμυντικό προπολογισμό σε ε, ευρωπαϊκό επίπεδο, ε, σε επίπεδο κράτους, ε, προέρχονται από το κεντρικό προπολογισμό από τους αμυντικούς προπολογισμούς. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν είχε νέες φιλοδοξίες ε, αυτές θα χρηματοδοτηθούν από τον προπολογισμό που ήδη υπάρχει για άλλους ε, σκοπούς. Εδώ και με την ΠΕΣΚΟ και με το Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο βλέπουμε ότι πρόκειται για νέο χρήμα που προέρχεται από τους κεντρικούς εθνικούς προπολογισμούς. Αν τα προσθέσει λοιπόν όλα μαζί κανείς, ε, είναι περισσότερα τα χρήματα που είναι διαθέσιμα για την άμυνα ε, θα έλεγα ότι είναι νέα χρήματα που πάνε σε υπάρχουσες προτεραιότητες ε, που έχουν ήδη εντοπίσει 22 κράτη με στη διάφορα διαδικασίες του ΝΑΤΟ. Εάν υπάρχουν ε, νέες προτεραιότητες που χρηματοδοτούνται από ήδη υπάρχοντα χρήματα, εκεί έχουμε άλλο ζήτημα. Κοιτάξτε, η πρόθεση είναι αυτή, είναι να υπάρχουν νέα χρήματα για υπάρχοντες στόχους. Τώρα για τις επιχειρήσεις. Ε, ρωτήσατε δύο πράγματα. Ποιος κάνει τι. Στη θέση μου πολιτικά δεν είναι σωστό να λέω ότι πρέπει να δούμε ποιος θα κάνει τι μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωση και ΝΑΤΟ, γιατί είναι σαν να λέει ένας οργανισμό στον άλλο τι πρέπει να κάνει, τι δεν πρέπει να κάνει. Σε έναν ιδανικό κόσμο, ναι, δεν θα έπρεπε να έχουμε παράλληλες ας πούμε αποστολές καταπολέμησης πειρατείας σε ένα μέρος του κόσμου ή οτιδήποτε παρεμφερές αλλά αφού δεν υπάρχει αυτός ο σαφής διαχωρισμός καθηκόντων και που δεν προβλέπεται άμεσα αυτό που μπορούμε να επιτύχουμε είναι να επιλύουμε τις ρήξεις στο το συντομότερο δυνατό. Όταν βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο όπως κάναμε στα Βαλκάνια πούμε, για δεκαετίες τότε θα πρέπει να διασφαλίζουμε τη σωστή επικοινωνία μεταξύ μας και να έχουμε επαφή, να ε, βελτιώνουμε τις προσπάθειες ενό του άλλου. Και στις περισσότερες περιπτώσεις είμαστε, το κάνουμε με επιτυχία. Κάτι άλλο ακόμα για τον κύριο Γκάλερ όσον αφορά την τυποποίηση, το ΝΑΤΟ εργάζεται εδώ και 60-70 χρόνια για την τυποποίηση και ακόμα δεν έχει φτάσει σε τέλειο σημείο, διότι πρόκειται μια προσπάθεια συντονισμού και συγχρονισμού εθνικών προσπαθειών πίσω από τις οποίες όμως δεν πάμε να υπάρχει εθνική κυριαρχία, οι εθνικοί σύμμαχοι που αποφασίζουν τι πρότυπα θέλουν και τι δεν θέλουν κτλ. Είναι μια συνεχής προσπάθεια και όπως υπενηχθήκατε κι εσείς θα ήταν πολύ καλό να είχατε δια πρότυπα η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη και χωρίς να δημιουργούν νέα πρότυπα που θα δημιουργήσουν νέα προβλήματα. Αυτά. Α δώσω το λόγο στον κύριο Διευθυντή. Thank you. Uh, so let me continue uh, trying not to repeat what uh, what Timo has already addressed, but but why not? why not? <laughs> Repetition is. Ε, θα ίσως χρειαστεί να επαναλάβω κάτι, άλλωστε η επανάληψη είναι η μητέρα της μάθησης. Ε, για το πρώτο θέμα, την αλλαγή της νοοτροπίας, της κουλτούρας. Ο Τίμορ ε, το εξήγησε με μεγάλη απλωτία γιατί συνεργασίες σε επίπεδο υπαλλήλων ε, γίνονται και πριν το 2014 και πριν την κοινή διακήρυξη της Βαρσοβίας. Φυσικά δίνει μια όθηση η διακήρυξη και ακόμα μεγαλύτερη όθηση θα έδινε η ύπαρξη διορατικών, οραματιστών πολιτικών και στις διοργανώσεις ε, με πολιτική βούληση να προωθήσουν το πρόγραμμα ε, ώστε να μην επικρατήσει η γραφειοκρατική προσέγγιση. Και φυσικά μας επηρέασε και το, το περιβάλλον, το τοπίο, ε, που ακριβώς λόγω της πίεσης ε, ε, προέκυψε επιτακτική ανάγκη να προσφέρουμε έργο και να δείξουμε αποτελέσματα. Οι υβριδικές απειλές και απειλές στον κυβερνοχώρο είναι πια πραγματικότητα. Το νιώθουν όλοι, νιώθουν το, το πόσο είναι η κατάσταση και η πίεση να εξασφαλιστεί προστασία και του κοινού. Και αυτή η πίεση έχει δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για την σημείωση άμεσης πρόοδου. Και χάρη και σε αυτή την πίεση συνεργάζονται πια οι διοργανώσεις. Επίσης κάτι που αποτελεί ίσως απόρρια ε, του προαναφερθέντος θέματος. Πριν από τρία χρόνια ανέλαβα το έργο μου και τότε ήταν τελείως διαφορετικό το τοπίο. Τότε τα θέματα της άμυνας, η συνεργασία με το ΝΑΤΟ ήταν ανήκουστο για την, Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η κατάσταση λοιπόν έχει αλλάξει ριζικά σήμερα. Και θα σας δώσω ένα αυτό παράδειγμα. Το ΝΑΤΟ με 2 εκατομμύρια ευρώ ε, στηρίζει ε, προγράμματα δημιουργίας ικανοτήτων, αμυντικών ικανοτήτων σε χώρες εταίρους. Γιατί φάνηκε ότι το ΝΑΤΟ ήταν ο καλύτερος φορέας εφαρμογής στον τομέα αυτό. Κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να συμβεί πριν από τρία χρόνια. Θα ήταν αδιανόητο. Έχει αλλάξει λοιπόν η προσέγγιση, η νοοτροπία, ο τρόπος με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εμπλέκεται σε θέματα ασφάλειας και άμυνας. Είναι ρηξικέλευτες αυτές οι αλλαγές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πιο φιλόδοξη πια, διεκδικεί ένα ρόλο, συμμετέχει στις συζητήσεις, διαδραματίζει ρόλο. Υπάρχει ορατή αλλαγή και θα πρέπει να αλλάξει πιο ριζικά και η Και το θέμα της ε, διακυβερνητικής προσέγγισης που συζητήσαμε και είναι και απαραίτητη, γιατί οι υβριδικές απειλές αποκαλούνται συχνά η σκοτεινή πλευρά της ε, σφαιρικής προσέγγισης και αν θέλουμε να έχουμε αποτελεσματική ανταπόκριση θα πρέπει ε, τα Υπουργεία να συνεργάζονται. Αν μείνει ο καθένας ε, στη γωνίτσα, δεν πρόκειται να σημειώσουμε πρόοδο. Και δεν είναι μόνο οι κυβερνήσεις απομονωμένες, γιατί μερικά πεδία, όπως το θέμα του κυβερνοχώρου, δεν είναι προνόμιο μόνο των κυβερνήσεων. Το 90% των δικτύων ε, ανήκουν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αυτές ουσιαστικά σχεδιάζουν το μέλλον στον κλάδο αυτό. Οπότε και αυτές ενέχονται και έχουν συμφέρον. Αν οι κυβερνήσεις θέλουν και δείξουν τη βούληση να λάβουν την, τις σωστές αποφάσεις σήμερα και να έχουν απήχηση και στο μέλλον, θα πρέπει ε, να συνεργαστούν και με τον ιδιωτικό κλάδο, με τις επιχειρήσεις αυτές. Θα πρέπει να αλλάξει τελείως... Ε, η νοοτροπία μας, γιατί οι απαιτήσει είναι σήμερα ριζικά διαφορετικές και θα πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Η αλλαγή της νοοτροπίας είναι πάντα το δυσκολότερο στοιχείο. Είναι ακόμη πιο δύσκολο από την κατανομή των πόρων η αλλαγή της νοοτροπίας. Και είναι και πιο χρονοβόρα διαδικασία, αλλά η πίεση αυξάνεται. Και άλλη λύση δεν υπάρχει. Σε ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών και μυστικών πληροφοριών. Όπως είπε και ο Τιμόρ, υπάρχουν κάποια προσκόμματα, υπάρχουν κάποια στενοπή προβλήματα. Το θέμα της ε, Κύπρου υπάρχει, δεν το έχουμε επιλύσει ακόμη και μέχρι ότου δοθεί λύση, οι περιορισμοί, οι μερικοί περιορισμοί θα παραμείνουν. Απλώς ε, ενισχύθηκε η πίεση προς τα κράτη-μέλη για να βρουν τρόπους να παρακάψουν κάποια προβλήματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα θεμελιώδη προσκόμματα έχουν αρθεί και πολύ συχνά ε, το ταυτίζουμε με το θέμα του το κυπριακό, αλλά δεν είναι τόσο περιορισμένο. Αν, ε, ε, ακόμη και αν αύριο λυθεί το κυπριακό, δεν είμαι σίγουρος ότι ως διαμαγές θα επιληθούν όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Αλλά σίγουρα η πίεση μας βοηθά, μας βοηθά να αναζητήσουμε πρακτικές λύσεις, όχι θεωρητικές, αλλά εύχριστες, έμπρακτες. Οπότε θα μας βοηθούσε σίγουρα η απρόσκοπτη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δύο οργανώσεων, αλλά αυτό εξαρτάται και από τα, αυτό εξαρτάται και από τα κράτη-μέλη. Ε, γιατί κάποια στοιχεία μπορούν και οι δύο να τα χρησιμοποιήσουν και να τα επεξεργαστούν. Υπάρχουν τρόποι λοιπόν για βελτίωση της κατάστασης και καλύτερα αποτελέσματα. Δεν διαβάζω εδώ τα γράμματά μου. Ε, για το σχόλιο για τις 42 προτάσεις. Όντως, μερικά θέματα τα, ε, τα λύσαμε ήδη, όπως το, η μονάδα Άλλα θέματα θα είναι ατέρμονα και θα χρήζουν συνεχούς επικαιροποίησεις και συμπλήρωσης. Και συνεχώς προτείνονται και νέες ιδέες. Όσο προχωρούμε στην υλοποίηση, όσο το απαιτούν από εμά οι περιστάσεις, θα εμπλουτίζουμε αυτόν τον κατάλογο. Το σημαντικό είναι να εξασφαλίσουμε μία ε, ιεράρχηση, γιατί σημαντικό κριτήριο είναι η προβολή, ε, το να είμαστε ορατοί. Κάτι κάνουμε στον τομέα αυτό το μήνυμα θα πρέπει να περνά στο ευρύ κοινό. Θα πρέπει το ευρύ κοινό να συνειδητοποιήσει ότι μένουμε συσφυρωμένοι και ενωμένοι και τότε έχουμε ε, αποτελέσματα, εν τη ενός ισχύς. Αυτό το αντιλαμβάνεται καλύτερα το ευρύ κοινό. Αν περιοριζόμαστε μόνο σε τεχνικά αποτελέσματα, θα είναι δυσνόητα για τον κόσμο. Θα πρέπει να παρουσιάσουμε τις επιτυχίες μας, θα πρέπει να δείξουμε ότι σημειώνουμε πρόοδο. σε ό,τι αφορά τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων ή των ευθυνών. Συμφωνώ με τον Τίμορ. Σε έναν ιδανικό κόσμο ε, μπορούμε να οριοθετούμε σαφώς τις αρμοδιότητες, αλλά κάτι τέτοιο είναι μόνο στη φαντασία μας. Και μερικές φορές, σε μερικούς τομείς, είναι θετική η ταυτόχρονη παρουσία και των διοργανώσεων. Στην Ουκρανία, για παράδειγμα, στα Δυτικά Βαλκάνια. Μερικές φορές η παράλληλη και ταυτόχρονη παρουσία είναι πιο επωφελής από την ε, παρουσία του ενός μόνο. Αλλά όχι πάντα. Αυτό που είναι σημαντικό όμως είναι να συνεργαζόμαστε ακόμη περισσότερο και να συγκρίνουμε τις προτάσεις μας και σε επίπεδο, σε φάση σχεδιασμού. Εκεί να άρουμε τη σύγκρουση αρμοδιοτήτων. Ήδη σε φάση σχεδιασμού. Οπότε οι συνεργάτες μου που ασχολούνται με το σχεδιασμό συνεργάζονται με τους ομολόγους του στο ΝΑΤΟ καθημερινά ώστε αν υπάρχουν παιδεία ε, με ταυτόχρονη παρουσία και των διοργανώσεων να συνεργαζόμαστε στο Ιράκ ή οπουδήποτε άλλο. Προτυποποίηση, προδιαγραφές, τυποποίηση, μακάρι. Μακάρι να το είχαμε, όπως μακάρι να έχουμε έναν ενιαίο φορτιστή ό,τι τηλέφωνο κινητό και χρησιμοποιούμε. Σίγουρα θα μας διευκόλυνε πολύ να έχουμε ενιαία πρότυπα. Να κρατήσουμε όμως αμύωτη την πίεση, ώστε ό,τι και αν κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα άμυνας, στο μέτρο του δυνατού να παρακολουθεί τις, τα μέχρι τώρα πρότυπα και τις προδιαγραφές, ώστε να μην έχουμε διαφορετικές δέσμες προτύπων και προδιαγραφών. Γιατί το ΝΑΤΟ τόσα από τα άλλα καθήκοντά του, ήταν και ένας οργανισμός ε, τυποποίησης. Οπότε θα πρέπει να αξιοποιούμε στο μέτρο αυτό το κεκτημένο του ΝΑΤΟ στην προτυποποίηση. Ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι όντως στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ε, κάποιους απομονωμένους θύλακες. Ε, ο καθένας δουλεύει στη γωνίτσα του. Αυτά θα πρέπει να τα ξεπεράσουμε και στην ανταλλαγή των πληροφοριών. Σε ό,τι αφορά την ανταπόκριση στις κρίσεις, έχουμε τρεις ξεχωριστούς μηχανισμούς για το Συμβούλιο, την ΕΕΔ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώς συνεργάζονται, άμα δεν ξέρουμε, ποτέ δεν επιδιώξαμε μια τέτοια συνεργασία. Τέτοιες ασκήσεις ε, CMX ε, δεν ξέρουμε πώς ε, λαμβάνουν χώρα και προσπαθούμε να έχουμε συνεργασία με τον ΝΑΤΟ και μερικές φορές δεν έχουμε καν συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε αυτή την άποψη είναι πολύ απαιτητικό αυτό το έργο. Τώρα, τι κάνουμε σε θέματα ασφάλειας και άμυνας. Καταρχήν, ε, ένα τμήμα είναι η συνολική προσπάθεια το Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ε, ε, εφαρμογή στην άμυνα της συνολικής στρατηγικής, το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράση για την Άμυνα, που προσπαθεί να δώσει κίνητρα για πρόοδο, δεν μπορούν να μείνουν ξεχωριστά από τη συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Δεν μπορούμε να τα διαχωρίσουμε. Είναι αλληλένδετα. Γιατί όλα αυτά δεν συμβαίνουν κενό. Πολύ σωστά το είπατε. Και μάλιστα, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτύχει στις προσπάθειές της να δημιουργήσει ικανότητες και να έχει περισσότερη επιχειρησιακή παραγωγή αποτελέσματα επιχειρησιακά. Αυτό δεν θα βοηθήσει μόνο την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας, αλλά θα βοηθήσει γενικώ την ολοκλήρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη και την, τον επιμερισμό των ευθυνών στο ΝΑΤΟ. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περισσότερε ικανότητε και μπορεί να έχει και αποτελέσματα σε συνεργασία με τον ΝΑΤΟ. Και το, το αντίστροφο ισχύει. Αν αποτύχουμε, τις ε, αρνητικές συνέπειες θα τις νιώσει και το ΝΑΤΟ και ε, θα φανούν και στην άλλη όχθη του Ατλαντικού. Έχουμε κοινά συμφέροντα και κοινή ευθύνη να φέρουμε σε αίσιο πέρα στο σχέδιο αυτό. Ρωτήσατε και για τον επιμερισμό των ευθυνών για θέματα κυβερνοασφάλεια μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Δύσκολο είναι να γίνει διαχωρισμό γιατί η αθεκτικότητα, γιατί περί αυτού πρόκειται σε τελική ανάλυση είναι εθνική ευθύνη πρώτα απ' όλα. Γι' αυτό θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τα μέλη μας, τα κράτη-μέλη, να επενδύουν και να συνεργάζονται για να, να ενισχύσουν την αθεκτικότητά τους και τις ικανότητές τους για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Πάντως, γενικώ η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο ικανή σε κανονιστικό επίπεδο, σε κανονιστικό πλαίσιο. Γιατί θεσπίζει οδηγίε που θα εφαρμοστούν παντού από τις κυβερνήσει, από τον κλάδο, τη βιομηχανία. Το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να το κάνει. Το ΝΑΤΟ έχει ένομες υποχρεώσεις να ε, υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να τηρήσουν τους κανόνες και τις οδηγίες. Αυτό το κάνουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΝΑΤΟ είναι πιο αποτελεσματικό στις επιχειρησιακές ικανότητες. Οπότε, από αυτήν την άποψη είναι καλό το όργανο που έχουμε. Ευχαριστώ κύριε Φιντά. Και ξέρω ότι κάποιοι συνάδελφοι θέλουν να λάβουν τον λόγο σύντομα, αλλά παρακαλώ πολύ σύντομα. Γιατί έχουμε και άλλο θέμα μετά με τους ομιλητές μας, με τον ομιλητή μας. Θα ακούσουμε λοιπόν πρώτα την Αναγκόμες, μετά τον Τζέφρι Φανόρτεν, Κύριε Ήκλοντε, σε αυτά τα πεδία που εντοπίζετε ευρωπαϊκή Ένωσης και ΝΑΤΟ θα μπορούσε να υπάρξει αυτή η συνεργασία, η διάρθρωση. Μετά την πτώση της Μοσούλης βλέπετε να αναπτύσσετε κάτι πια τέτοια δυνατότητα για το Ιράκ. Εγώ θα προτιμούσα και πριν ακόμη, αλλά οπωσδήποτε τώρα. Κύριε Σβανόρτεν. Μα η προηγούμενη μου ερώτηση δεν απαντήθηκε. Δεν απαντήθηκε. Πώς βλέπετε το μέλλον ε, των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit ε, στο χώρο της άμυνας. Παρακαλώ. Ναι, επιτρέψτε μου να απαντήσω πρώτος. Είναι πολιτικό θέμα το Brexit. Είναι θέμα διαπραγματεύσεων. Δεν έχω κανένα, καμιά κρυστάλλινη μπάλα για να το διαβάσω το μέλλον. Για τη διάρθρωση βεβαίως είναι πολύ περίπλοκες οι διαπραγματεύσεις. Δεν ξέρω πώς θα προχωρήσουν. Λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να καταλάβουν όλα τα στοιχεία του μοσαϊκού αυτού, του ενίγματος αυτού. Δεν είμαι αρκετά ικανός εγώ. Ιράκ. Το να το ίδιο μπλέκεται. Έχει ίδια ομάδα εκεί η αποστολή. Εμείς ε, είμαστε στην ε, διαδικασία της εκείνης της διαδικασίας ε, πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Επομένως, αναπτύσσεται άλλος ένας χώρος δραστηριοτήτων, επιχειρήσεων, ένα πεδίο επιχειρήσεων και εδώ έχουμε πάρα πολύ στενό συντονισμό. για να έχουμε μόνο συμπληρωματικότητα και όχι σύγκρουση ασυμβατότητα. Και η Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο ομιλητάς για την ε, επίκαιρη, εύθετη και διεξοδική κάλυψη του θέματος. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση και είμαι βεβαία πως θα επανέλθουμε συντομότατα. Sorry Συγγνώμη για αυτή το διάλειμμα χρειάστηκε να πάρω κάποιο φάρμακο γιατί φαίνεται να είναι κολλητική, κολλητικός ο βήχας εδώ. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε λοιπόν το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης με θέμα περί την περιφερειοποίηση των αποστολών της κοινή πολιτικής ασφαλείας και άμυνας στην περιοχή του Σαχέλ και ανασκόπηση από την εμπειρία της EUTM στο Μαλί που δραστηριοποιούμαστε εδώ και αρκετό καιρό με την αποστολή αυτή στο Μάλι Εξακολουθούμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και θα την παρακολουθούμε και στις επόμενες ε, συναντήσεις της ε, ΣΕΝΤΕ, της εξελίξης εκεί. Να σας παρουσιάσω τον αξιότιμο μιλητή. Είναι προϊστάμενος του τμήματος ε, της ΕΕΔ, ασχολείται με τον σχεδιασμό και ειδικότερα με την ανάπτυξη της θεσμικής μας παρουσίας ε, στην περιοχή του Σαχέλ. Σας παρουσιάζω λοιπόν τον κύριο Ζακ Φχαντά, που είναι απευθείας αρμόδιος γι' αυτό. Προκείται για το τελευταίο σημείο. Είναι το τελευταίο λοιπόν σημείο της ημερήσιας διάταξης. και πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Δεν τελειώνει εδώ η δέσμευση της ΕΝΤΕ, όμως την επόμενη Δευτέρα ξεκινάμε την αποστολή στην Νάπολη, στην Κατάνια και στην Μεσόγειο. για να δούμε τις ε, δράσεις της ε, κοινής ε, τις ασφάλειες και άμυνας εκεί. Έχετε το λόγο, κύριε Φράντα. Ευχαριστώ πολύ, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων. Ζητά συγγνώμη, πρόεδρος για τον τρόπο τον οποίο πρόφερε το όνομα του ομιλητή. Συμβαίνει, κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, ονομάζομαι Ζακ Φράντα. Προέρχομαι την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, στη Διευθύνση Σχεδιασμού ε, Διαχείρισης Κρίσεων. Ευχαριστώ που με καλέσετε σήμερα για να δούμε την κατάσταση σχεδόν ένα χρόνο μετά από την τελευταία μου παρουσία εδώ. Είναι σαν μια επέτειος λοιπόν εδώ στο Κοινοβούλιο μετά από την επίσκεψή σα στο Μάλι. Ε, τρία πράγματα θα έπρεπε να παρουσιάσουμε. την περιφερειοποίηση που βρισκόμαστε, στην παρουσίαση θα συμπεριλάβω την G5 Sahel, πόσο έχουμε μπλακεί, ε, πώς έχει γίνει αυτή η περιφερειακή δράση και θα τελειώσω με την EUTM. Θα κάνω μια ομιλία αρκετά συνοπτική και θα είμαι έτοιμος να απαντήσω στις ερωτήσεις σας στη συνέχεια. Η δράση λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σαχέλ και ειδικότερα στο Μάλι είναι καθοριστική. Όλοι γνωρίζουμε τις, ε, το πώς ξεκίνησαν τα πράγματα και πώς έχει το περιβάλλον σήμερα. Εδώ και ένα χρόνο, από τότε που ήρθα να σας μιλήσω πριν από ένα χρόνο για την περιφερειοποίηση, τα πράγματα έχουν αλλάξει από άψη ασφάλειας. Δεν έχει αποδυναμωθεί μεν η απειλή. Θα έλεγα ότι έχει αποδυναμωθεί το κέντρο του Μάλι η δράση των διεθνών εταίρων των Ηνωμένων Εθνών, της Γαλλίας, ε, ε, μέσα της Μαρκάν και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα των δύο αποστολών που έχουν παρουσία στο Μάλι και τα άλλα προγράμματα που υλοποιήθηκαν ε, δείχνουν πόσο δεσμευμένη είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χώρα αυτή αλλά και για την περιφέρεια. Όσον αφορά την περιφερειοποίηση, όταν σας παρουσίασα την κατάσταση όπως είχε πριν από 10 μήνες, Βρισκόμασταν στη φάση έγκρισης από τα κράτη-μέλη έκτοτε. Ξεκίνησε η διαδικασία, την οποία θα σας περιγράψω με τρόπο απλό. Η πρώτη φάση συνίσταται στην υλοποίηση ενός δικτύου ασφαλείας σε πέντε χώρες του Ισαχέλ, Μαυριτανία, Νίγηρας, Τσάντ, Μπουρκίνα Φάσο, Νίγηρας, το ξανά λέει ο και Μάλι. Φαίνεται φιλόδοξο αυτό που σας περιγράφω, αλλά θα δείτε ότι αντιστοιχεί στην επόμενη φάση, σε μια ενισχυμένη φάση, ε, σε σχέση με τις ε, προσδοκίες ε, για το σύνολο της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σαχέλ. Σε αυτή τη φάση υπαριθμών 1 έχουμε δύο αξιωματικούς ασφαλείας ή άμυνας ανά στι στις χώρες που ανέφερα, εκτός από το Μάλιο, που υπάρχουν ήδη αποστολές, οι οποίοι θα συμβάλλουν στη δικτύωση στη δημιουργία ενός δικτύων που θα τροφοδοτήσουν τους θεσμούς με μια σειρά αξιολογήσεων σε σχέση με το πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να σας υπενθυμίσω ότι τρεις προτεραιότητες που έχουμε για αυτή την περιφερειοποίηση είναι η υποστήριξη της διασυνορικής συνεργασίας του Σαχέλ, η υποστήριξη των δομών περιφερειακής συνεργασίας και ειδικότερα των χωρών του G5 του Σαχέλ και εκεί η ενίσχυση των εθνικών ικανοτήτων των πέντε χωρών αυτών. Εμείς ε, εδώ βοηθάμε σε περιφερειακές δράσεις, ε, διακρατικές, είτε συλλογικές, είτε μεταξύ ορισμένων κρατών μελών από αυτές τις χώρες. Γι' αυτό όταν λέω για το G5 θα το καταλάβετε καλύτερα. Όσον αφορά τους εμπειρογνώμονες ε, στην αποστολή ΚΑΠ 5 Μαλή θα έχουμε ε, ένα κέντρο που θα ασχολείται με τη συλλογή των πληροφοριών, την ανάλυση τους, την αποστολή τους στις Βρυξέλλες. Θεωρούμε στις αρχές του 2018 να υπάρχει αυτό που ονομάζουμε need assessment αξιολόγηση αναγκών και κενών ε, σε σχέση με τις ικανότητες που σας περιέγραψα. Οι δράσει δηλαδή δεν εστιάζονται μόνο στις χώρες. Αυτό το περιφερειακό σχέδιο δράσης στη συνέχεια θα συζητείται μεταξύ κρατών μελών εδώ και θα αποφασίζετε ποιες δράσεις θα γίνουν στο μέλλον σε κάθε μία από αυτές τις χώρες σε ποιο πλαίσιο ε, κατάρτισης, με ποιο δυναμικό και με ποιο χρονοδιάγραμμα. Και μετά θα δούμε τους αξιωματικούς επαφές ε, που θα διασφαλίζουν ότι ε, ό,τι υλοποιείται δεν θα χαθεί. Οι χαμηλές επενδύσεις σε κατάρτιση σε ορισμένες χώρες ε, ε υπάρχουν κενά σε προσωπικό, δεν, Θέλουμε να καταρτίζουμε τον κόσμο ώστε να δημιουργούμε ικανότητε δυνατότητε ε, που να βοηθούν του πάντε και ειδικότερα τι χώρε που συμμετέχουν οικονομικά. Εκεί λοιπόν σε πρώτη φάση θα γίνεται μια συλλογή των πληροφοριών, αξιολόγηση των κενών και των αναγκών και εκεί θα αποφασίζετε ποιε δράσει πρέπει να τους ε, να δημιουργήσουμε για αυτού για τη φάση 2. Η φάση 2 θα γίνει τέλη του 2018, έγκριση από τα κράτη-μέλη, όπου θα αποφασιστεί πώ θα διεξαχθούν οι δράσει. Εδερχόμαστε και σε αυτό που είπε ο διευθυντή μου προλίγου, το η σύνδεση μεταξύ ασφάλεια και ανάπτυξη, που κατά την άποψή μου θα βασιστεί και σε ε, ανάγκε ε, που μπορούμε να καλύψουμε με δράση μας σε αυτές τις χώρες. Στη φάση αριθμός 2, στην περιφερειοποίηση, τα πράγματα μπορούν να πάνε πιο γρήγορα. Διότι πρόσφατα είδαμε να επισέρχεται ένα νέο παράγοντα. Κάτι που έδειξε ότι ήμασταν ε, πολύ καλές οι προβλέψει μας στην αξιολόγηση των αναγκών ε, τη περιοχή. Και εδώ έρχομαι στο δεύτερο σημείο. Η G5 δημιούργησε μία δύναμη, τη δύναμη G5, που ψηφίστηκε στις 27 Ιουνίου ε, στα Ηνωμένα Έθνη στο ψήφισμα 2359 πολύ σημαντικό διότι ευθυγραμμίζει τις προσπάθειες για την ενδεχόμενη διεθνή στήριξη αυτής της δύναμης. Ποια είναι αυτή η δύναμη, η G5 λοιπόν. Ε, είναι μια δύναμη όπου οι πέντε χώρες της ε, περιοχής που ανέφερα συντονίζουν τις δυνάμεις τους για μια συλλογική δράση ε, αντιμετώπισης συλλογικών απειλών. Μιλάμε για μια δύναμη περίπου 5.000 ατόμων και ένα μη στρατιωτικό σκέλο ε, για τη χωροφυλακή ε, που χωρίζεται σε τρει άξονε. Ανατολικό άξονα, ε, Μαυριτανία και τα στο κέντρο, Μάλι, Μπουρκινα και Νίγηρα και δυτικά στο Τσάντ. Πού βρισκόμαστε σήμερα. Έχουμε μία δύναμη που εγκαθίσταται στο κεντρικό σκέλος θα είναι μια διαστρατητική ομάδα στο Μάλι που θα συντονίζει μια δύναμη η οποία θα αναπτυχθεί στην Πουρκίνα, στην Ήγερα και στο Μάλι. Εδώ συγκεντρώνονται πολλές δυνάμεις, πολλές πρωτοβουλίες ε, γαλλογερμανικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα το έχετε ακούσει, διότι αποφασίστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση να χορηγήσει 50 εκατομμύρια ε, για αυτή τη δύναμη. Όλα αυτά, διότι όπως εξήγησα στην αρχή, η κατάσταση της ασφάλειας υποβαθμίζεται στο κέντρο, στο κέντρο του Μαλή και δεν υπάρχουν αρκετά μέσα για την αντιμετώπιση και την ανάσχεση των απειλών που βλέπουμε. Δεν μιλάμε για την εκρίζωση των θυλάκων, αλλά για τον έλεγχο της κατάστασης. Και εκεί οι προτεραιότητες της G5 όπου θα χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή που μπορούν να, με τα οποία μπορούν να συμβάλλουν οι άλλε χώρε. Μιλάμε για αντιμετώπιση τη τρομοκρατίας, τη διακίνηση ναρκωτικών και ανθρώπων, ε, της αυθαιρεσίας των κρατών, να διευκολύνουμε τι ανθρωπιστικέ δράσει και να συμβάλλουμε στην υλοποίηση των δράσεων για την ανάπτυξη των χωρών του Σαχέλ. Είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλή στρατιωτική δράση. Ε, με ένα χρονοδιάγραμμα εξαιρετικά ευρύ, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αδράξει την ευκαιρία να αναλάβει την πρωτοβουλία. Ε, ε, μέχρι το τέλος του έτους θα απαιτηθεί μεγάλη βοήθεια, αλλά δεν θα αρκέσει. Για να κλείσω την παρουσίασή μου, να σας ε, μιλήσω για την EUTM και το ρόλο των ε, αποστολών ε, πολιτικής ασφάλειας και άμενας. Έχουμε δύο μη στρατιωτικέ αποστολέ στον Νίγηρα και στο Μάλι και μη στρατιωτική αποστολή την EUTM Μάλι. Οι δύο μη στρατιωτικέ αποστολέ μπορούν να καταρτήσουν τους εμπειρογνώμονες ε, στις δυνατότητε που εργάσαν προηγουμένως, ε, την πλησίωση ώστε να αναπτυχθούν οι σωστές πρακτικές και μέθοδοι για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της του οργανωμένου εγκλήματος ε, και παράλληλα να φροντίσουν τα προβλήματα να μένουν εκεί, να μην εξαχθούν. Και εκεί να υπερασπιστούμε τους στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης, να υπάρχει μια σταθερότητα δηλαδή η οποία θα επιβληθεί εκεί, από την οποία θα επωφεληθούμε και εμείς και μετά θα ακολουθήσει η φάση 2 της περιφερειοποίησης και όσον αφορά την UTM θα υπάρξει μια σημαντική δράση, είναι η πρώτη στρατιωτική δράση που υπάρχει εκεί, η πρώτη στρατιωτική αποστολή η οποία έχει αρχίσει ήδη να βοηθά με τη σύνταξη εγγράφων ε, επιχειρησιακών σχεδίων, έτσι τα ονομάζουμε το επιτελείο που θα εγκατασταθεί στο τη Σεβαρέ, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Μάλι. Το Προεδρείο τη G5, όπω είπα σήμερα, ε, το έχει το Μάλι και στη συνέχεια θα ε, προσφερθούν καταρτήσει Στο πλαίσιο που περιέγραψα το EUTM Μάλι, όπω είπα, έχει μια νέα εντολή. Οι δύο πρώτε εντολές ήταν για τη δημιουργία στρατιωτικών δυνάμεων του Μάλι, αλλά εκεί ξεχάσαμε τι σημαίνει αποστολή ε, κοινή πολιτική άμυνα και ασφάλεια. Υπάρχουν τρει πυλώνες. Πρώτο, ε, πυλώνα στρατηγικό, βοηθάμε την κυβέρνηση ε, στην καλύτερη υποστήριξη και οργάνωση των στρατιωτικών δυνάμεων. Μετά έχουμε τον πυλώνα κατάρτισης που ασχολείται με το προσωπικό και μετά ε, ένα άλλο πυλώνας εκπαίδευση πιο ορατό, που πρέπει να ειδωθεί όμω μαζί με του δύο άλλου. Για την εκπαίδευση λοιπόν στην πρώτη εντολή οκτώ μάχημες μονάδες εκπαιδεύτηκαν στο Μάλι που είναι έτοιμες σήμερα το τάγματα έχουμε ε, εγκαταστήσει αυτές τις ομάδες ε, στο Κορεκορόμ στο Πολυκορόμ για να υπάρχει μια ε, αποκέντρωση. Έχουμε στο Σεγκού, στον Καό και σε άλλο σημεία και έτσι μπορούμε ευκολότερα να πάμε σε διάφορες περιοχές του Μάλι και να βοηθήσουμε στην επίλυση ζητημάτων και στις αποστολές στις περιφέρειες του Μάλι. Θα μου πείτε ποτέ δεν, αρκεί για να καλύπ... δεν αρκούν όλα αυτά για να καλύψουν τις ανάγκες, αλλά έχουμε το στρατό του Μάλι που μας βοηθά, που είναι καλός εταίρος, έχει απώλειες και που μόλις στρατολόγησε 5.000 άτομα η UTM Μαμάλη βοήθησε και στην ξεφνική απροσδόκητη ε, εκπαίδευση. Έχουμε καταρτήσει λοιπόν τους εκπαιδευτές για αυτά τα νέα τάγματα. Ε, μια αποστολή που εξετελέσει με μεγάλη επιτυχία και ταυτόχρονα συνεχίζουμε με το στρατηγικό πυλώνα και τον πυλώνα της εκπαίδευσης. Θα αναθεωρήσουμε την εντολή αυτής της αποστολής πριν τα τέλη του έτους και θα σχεδιάσουμε τη μελλοντική εντολή βάσει τη εξέλιξη τη περιφερειοποίηση και του G5 και βάσει και των προτεραιοτήτων. Γι' αυτή είναι και η βούληση των κρατών μελών. Όλε αυτέ οι αποστολέ ε, δεν πρέπει να έχουν μια εντολή που να σχετίζεται μόνο με τη δράση και το κέρδο τη χώρα. Όλα πρέπει να γίνονται σε περιφερειακό επίπεδο διατηρώντας τη βασική εντολή αυτή των αποστολών. Κάτι τελευταίο που θέλω να προσφέρω, να, να παρουσιάσω, συγγνώμη. Θα έχετε ακούσει για την επίθεση του 18 Ιουνίου στον Παμάκο όπου ένας στρατιώτης δυστυχώς του UTM έχασε τη ζωή του και θέλω να εκφράσω τα μου προς τον Πορτογαλία διότι ο λόγος στρατιώτης ήταν Πορτογάλος αποκομίζουμε τα διδάγματα αλλά όταν μιλάμε για αποτελέσματα των αποστολών UTM ε, των αποστολών στο Μάλι, ε, σε τέτοια, από τέτοια περιστατικά μαθαίνουμε πράγματα αυτός ο άνθρωπος σε δύο χρόνια θα έχει... Οι αστυνομικοί του Μαλή βοήθησαν και οι δύο αποστολές συνέβαλαν ε, για να βοηθήσουν το στρατό ε, και έτσι αποκομίσαμε διδάγματα για να συνεχιστεί αυτός ο ενάρετος κύκλος βοήθειας των δράσεων ενημέρωσης, ε, βελτίωσης της δράσης μας. Εδώ θα κλείσω. Αυτό το γεγονός δείχνει ότι από τότε που έχουμε παρουσία στο Σαχέλ και στο Μάλι, παρότι είναι αργή η πρόοδος, μην ξεχνάτε ότι έχουμε να κάνουμε χώρε χώρες σε κρίση, ε, σε εμπόλεμη κατάσταση. Η δράση μας λοιπόν παρόλα αυτά ε, έχει αποτελέσματα, αν και αποδυναμωμένα σε σχέση, λόγω των περιορισμών, αλλά είναι αποτελεσματική. Σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σα για να απαντήσω στι ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά. Ποιο θέλει το λόγο παρακαλώ, ο κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ. Και βεβαίω Ναι, περιμένω. Εύχομαι για μας και για το μαλλί πάνω απ' όλα, να ευοδοθούν αυτές οι προσπάθειες και έξω και την... και να καθίσταται αντιληπτή η ύπαρξη του κράτους και έξω από την πρωτεύουσα. Αυτό μπορούμε εμείς να προσφέρουμε είναι η ευρύτερη περιοχή να αποκτήσει τις απαραίτητε δομές ώστε να μπορούν μόνοι τους οι Αφρικανοί να επιτύχουν τους στόχους αυτούς. Εσείς πιστεύετε ότι στον τομέα ΕΚΟΒΑΣ και γενικά τη συνεργασία μεταξύ αυτών των ε, πέντε κρατών μπορούμε να διαγνώσουμε μια μόνιμη πολιτική βούληση ενδεχομένως και για αυτοχρηματοδότηση. Γιατί πρέπει κάπου να έχουν τη διάθεση και αυτοί να σταθούν στα πόδια τους μόνοι τους. Βλέπετε κάποια τέτοια τάση. Η κυρία Γκόμες. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον κύριο Φράντα γιατί και εσείς και η κυρία Μογκερίνη της προάλλες εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους για, την, για το θάνατο του Πορτογάλου στρατιώτη που έχασε τη ζωή του με την επίθεση στην στρατιωτική αποστολή μας στο Μαλί. κατάλαβα την προσπάθεια συνδυασμού των ε, επιχειρήσεων και με τις επιχειρήσεις μας στις άλλες χώρες της περιοχής. Ε, είναι απαραίτητη αυτή η συνεργασία για να ε, αντιταχθούμε στις τρομοκρατικές ενέργειες και στην τρομοκρατία γενικώ που λιμένεται την περιοχή. Τι γίνεται όμως με την στρατιωτική εκπαίδευση και θεωρείτε ότι συμμετέχετε και λαμβάνετε την ε, δέουσα υποστήριξη σε μια, μια πιο μακρό προσπάθεια που στόχο έχει την ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης αλλά ίσως και την ενίσχυση ακόμη και της ανάπτυξης γιατί γνωρίζουμε ότι αυτή είναι η αιτία των συγκρούσεων και δίνει προσχήματα και κάνει τους ε, ανθρώπους πιο ευάλωτους ε, στη ρητορική των τρομοκρατικών ομάδων και έτσι στρατολογούν πιο εύκολα. Γιατί ε, έχουμε αναπτύξει τεράστια στρατητικά μέσα που έδωσαν και καρπούς ε, σε ό,τι αφορά την αντίδραση των ενόπλων δυνάμεων εκεί. Αν όμως σε επίπεδο ανάπτυξης και διακυβέρνησης δεν βελτιώνεται η κατάσταση και δεν ε, διαπιστώνουν την βελτίωση οι ντόπιοι, ό,τι η στρατιωτική προσπάθεια και να έχουμε δεν θα αποφέρει Πως απλώς θα μας εκθέτει ακόμη και περισσότερο, θα μας κάνει πιο ευάλωτου. Θεωρείτε ότι η στρατιωτική αυτή αποστολή ε, πλαισιώνεται δεόντως από αντίστοιχε προσπάθειες σε ανάπτυξη και διακυβέρνηση. Ο κύριος Έθριτς, συνεχίζοντας τη τελευταία ερώτηση, με ενδιαφέρει η συνάρθρωση αυτών των δυνάμεων και η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αποστολών και αντιλαμβάνομαι την σταδιακή προσπάθεια που γίνεται και την προοδευτική και χαίρομαι. Ε, διερωτώ με όμως ε, ποια είναι τα όρια αυτής της εμπλοκής, ε, της ανάμιξης. Επειδή υπάρχουν ε, πολλές επιπλοκές και αλλοδαπή παράγοντες, πρόκειται για μια περιοχή χαοτική, ε, και μιλήσαμε για τις θλιβερές απώλειες κάποιο μελών της αποστολής. Ε, ποιο, ποιος είναι ο κίνδυνος αυτής της ε, αποστολής, γιατί πολύ συχνά η Δύση είναι πλάκη σε συγκρούσεις για πολλούς και διάφορους λόγους, προσπαθώντας να ενισχύσει την παρουσία του σε μια περιοχή, αγνώντας μερικές φορές το τελικό σημείο και ε, χωρίς να δίνει τη δέουσα έμφαση στον τρόπο παραπατρισμού αυτών των στρατευμάτων μας. Ε, ε, ποιος είναι ο κίνδυνος τέτοιων αποστολών. Ε, γιατί πολύ φοβάμαι ότι θα, θα, θα συνεχίσετε να υφίσταται τις συνέπειες ε, των καταλήπων του απεικιοκρατικού παρελθόντος και δεν θα αποφεύγουμε μερικές καθημερινές τραγωδίες. Ευχαριστώ. Δεν ζήτησε άλλος κανείς το λόγο. Θα ήθελα τώρα και εγώ να θέσω μια ερώτηση, μάλλον δύο. Η γενικότερη περιοχή ε, είναι όντως ε, έκριθμη. μερικές φορές. Ε, και τις συνέπειες αυτής της ε, διέλευσης του μεταναστευτικού κύματος προς την Ευρώπη και παρά τις συντονισμένες ε, προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τα σχόλια όταν μιλούμε για την γαλλική παρουσία στον Ήγηρα ή τη συνεργασία ε, των Αμερικανών και την Αμερικανική συνεισφορά. Είναι δυνατόν ή εύκολο και ποια είναι η προστιθέμενη αξία πιθανού συντονισμού και ποιοι είναι οι τρόποι συντονισμού της παρουσίας και των ενεργειών των διαφόρων παραγόντων που βρίσκονται στην περιοχή. Εμείς διαπιστώσαμε ότι ήταν πολύ χρήσιμη η παρουσία της Γαλλίας στην περιοχή ε, και η Γαλλική Συνιστόσα ήταν πολύ πεπειραμένη, ε, με μεγάλη βούληση ε, ανάμεξης και με πολύ θετικά αποτελέσματα και σε άλλους τομείς. Ερωτώ λοιπόν τι δυνατότητες υπάρχουν για συντονισμό των προσπαθειών και των ενεργειών σε περίπτωση που παρίστανται περισσότεροι παράγοντες. Ε, επίσης, είχαμε πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις στον Πατακλάν, στο Παρίσι και αλλού και η Γαλλία μετά από αυτό ζήτησε μια βοήθεια ε, για να παρασχεθεί μια ενίσχυση στις δικές προσπάθειες σταθεροποίησης της περιοχής του Σαχέλ. Υπάρχει μια συλλογική ανταπόκριση σε αυτό το αίτημα της Γαλλίας για να μειωθεί κάπως η δική της παρουσία εκεί. Η μονοδημέρης ήταν αυτή η αίτηση της Γαλλίας προς μεμονωμένες χώρες. Πώς εκτιμάτε γενικώ τη συνολική παρουσία του δυτικού κόσμου και χωρών μελών του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Και πώς αξιολογείται τα αποτελέσματα αυτής της παρουσίας. Μιλήσαμε πριν και για την εντολή της στρατιωτικής μας αποστολής στο Μαλί και τη... μιλήσαμε για την εντολή και άλλων αποστολών στην περιοχή. Ποιο κατά τη γνώμη σας είναι το χρονοδιάγραμμα, ο χρονικός ορίζοντας της παρουσίας μας ε, εκεί. Έχετε το λόγο, δεν ξέρω αν θα ακολουθήσει και δεύτερος γύρος προς το παρόν. Σας ακούμε. Σας ευχαριστώ πολύ, εύστοχες οι ερωτήσεις σας ε, και οξυδερκείς δείχνουν ότι είστε εξοικειωμένοι με το αντικείμενο, ε, κάτι που με χαροποιεί και πραγματικά βάζετε το δάκτυλο επί των τύπων των ήλων. Μας χτυπάτε στον κάλο κατά κάποιο τρόπο. Θα προσπαθήσω να απαντήσω κάπως γενικά, καταρχήν απαντώντα στη δική σας ερώτηση, κυρία Πρόεδρε, για τις κοινέ προσπάθειες, τα συμφέροντά μας και γιατί έχουμε εμπλακεί στο Σαχέλ. Καταρχήν για τις σταθεροποίηση της περιοχής και ε, για δικούς μας λόγους, για τη μετανάστευση, για τη δρομοκρατία, για τη γάγκρενα που συνιστούν αυτές ε, οι ομάδες ε, τύπου Μποκοχαράμ, Ισλαμικού κράτους, που είναι μάστιγα και για την Αφρικανική Ήπειρο και με τις ε, αποστολές της ΚΠΑ και με άλλα μέσα. Έχουμε βοηθήσει την πολυεθνική δύναμη ε, της Αφρικής στο Τσάντ, για παράδειγμα. Έχουμε την δύναμη του G5 στο Σαχέλ. Βοηθάμε τους Αφρικανούς, αλλά ταυτόχρονα ευλογούμε και τα γένια μας, γιατί έχουμε και τα δικά μας συμφέροντα εκεί. Επίσης, ό,τι αφορά τη διεθνή συνεργασία, έχουμε διάφορους παράγοντες, καταρχήν διμερούς χαρακτήρα όπως η Γαλλία, η ε, η Αμερική και έχουμε και κάποιες δράσεις ε, ε, αντιτρομοκρατικές ε, που γίνονται όταν κανένας δεν τις αναλαμβάνει ουσιαστικά του πάντματος, του φάσματος. Τώρα στο Μάλι έχουμε τη Μίνωσμα που έχει συμμετέχει και στη συμφωνία του, του, του Αλιγερίου και φυσικά προσπαθούμε να αποφύγουμε τις επικαλύψεις. Και τρίτος παράγοντας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που δραστηριοποιείται περίπου στο ίδιο πεδίο, είτε στο στρατιωτικό είτε στο μη στρατιωτικό, με την αποστολή δημιουργίας ικανοτήτων. Και εμεί με την EU-CAP προσπαθούμε ακριβώ να δημιουργήσουμε ικανότητε. Ενώ η UTM είναι στρατιωτική αποστολή, εκπαιδεύει ενόπλε δυνάμει. Και Αντικείμενο του συντονισμού είναι να αποφύγουμε τις επικαλύψεις, την επανάληψη των προσπαθειών, πρώτον, και δεύτερον, να εξασφαλίσουμε μια συμπληρωματικότητα των δράσεων. Αυτό είναι το συζητούμενο διαρκώς και περίπλοκο βέβαια και επίσης να κάνουμε κάτι που δεν κάνουν άλλοι. Και εδώ σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών προσπαθούμε να κάνουμε ότι δεν κάνουν οι υπόλοιποι παράγοντες στο Μάλι. Και έχουμε ένα κινούμενο στόχο, κάτι που είναι δύσκολο γιατί οι παράγοντες από το Μάλι σε θα επανέλθω σε λίγο στο πολιτικό ερώτημα της κυρίας Γκόμες, οι πολιτικοί παράγοντες στο Μάλι είναι πολύ εργοκίνητοι μερικές φορές ε, σε πολιτικό επίπεδο και δεν μπορούμε εμείς να υπακοτασταθούμε στο έργο τους. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις, τους πολιτικούς ηθήνοντες του Μάλι ώστε να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Εμείς μόνο βοήθεια μπορούμε να δώσουμε, μία απλή συμβολή. Το λιθαράκι μας βάζουμε στο οικοδόμημα, δεν μπορούμε να το κατασκευάσουμε όμως εκ Μετά τις επιθέσεις στις θερμοκρατικές στο Παρίσι, η Γαλλία ψήφισε το άρθρο 42.7, δηλαδή ενίσχυσε ε, την συμμετοχή της στη Μίνουσμα. Ένα από τα, μια από τις αδυναμίες της Μίνουσμα είναι ότι η ικανότητα διοίκησης και ελέγχου και η επιμελητιακή ικανότητα και η ικανότητα άμεσης δράσης ε, ήταν κάπως προβληματική. Οπότε ε, η Γαλλία πρόσφερε στη Μίνουσμα με τα, τις ικανότητές της, την πείρα της και μετά συμμετείχε και η Γερμανία και άλλες χώρες και έτσι ε, ενισχύθηκε η Μίνουσμα που είναι η στρατιωτική αποστολή των ΗΠΑ που έχει τις μεγαλύτερες απώλειες τα τελευταία χρόνια. Οπότε και για τη Μίνουσμα, την αποστολή αυτή του η πρόκληση είναι μεγάλη. Επίσης, ε, τι εντολή αναθέτουμε σε τέτοιες αποστολές του ΟΗΕ σε σχέση με τα λίγα μέσα που έχει στη διάθεσή της μια τέτοια αποστολή. Χρειάζεται λοιπόν συμπληρωματικότητα και συντονισμός και φυσικά και μία συνέχεια. Κύριε Έθριτς, ε, το Mission Creep που είπατε, δηλαδή μία αποστολή που διονύζεται, είδαμε τι συνέβη ε, και σε άλλες χώρες και διάσημα παραδείγματα, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δική μας αποστολή και πάει πιο παλιά είναι στη Βοσνία. Ε, σε ε, πολύ μικρή σε σχέση με τη Φινούλη, με άλλες του ΟΗΕ που ήταν με 30.000 προσωπικό. Και αυτό θέλουμε να απεφύγουμε, να διαονίζονται οι, οι αποστολές μας. Γι' αυτό και έχουμε τακτικά αξιολογήσει με τα κράτη-μέλη που αποφασίζουν για τη χορήγηση του προσωπικού. Γιατί αν η εντολή δεν εξυπηρετεί τα κράτη-μέλη, δεν στέλνουν πια προσωπικό. Και αυτή είναι η ασφαλιστική δικλίδα για να μην διονύζονται οι αποστολέ μα. Πάντω όλε μα τι αποστολέ ε, ε, δεν είναι στατικές, είναι δυναμικές και ευέλικτες. Και Φυσικά σκεφτόμαστε και το μέλλον, το αύριο, την επόμενη φάση και προσαρμοζόμαστε στις αποστολές. Και η ικανότητα απορρόφησης ε, και το local buying που λέμε, η ανάληψη ευθυνών σε τοπικό επίπεδο για μας έχει κέρια σημασία και γι' αυτό διαμορφώνουμε και τις αποστολές μας για να αποφύγουμε να διαονίζονται οι ε, αποστολές μας. Και μάλιστα κλείσαμε δύο τέτοιε αποστολέ, στο Κογκό, στην Κινσάσα, μία αποστολή στη Γουινέα Μπισάου. Και τα κράτη-μέλη αποφασίζουν αν παρατείνουν ή όχι μια, την εντολή μιας αποστολής. Υπάρχει έλεγχος της ποιότητας που εξασφαλίζεται από τα κράτη-μέλη. Στο, στο θέμα του Μαλή, φυσικά υπάρχει ένα όριο με βάση τη, την εντολή του, του, της ΚΠΑ εμείς ε, δεν συμμετέχουμε στις μάχες, απλώς εκπαιδεύουμε τις ένοπλες δυνάμεις και βλέπουμε ε, τα αποτελέσματα. Και κάποια στιγμή ε, διαπιστώνουμε προβλήματα εξοπλισμού, για παράδειγμα, ή στήριξης. Και αυτό είναι και το διακύβευμα. Και αυτό επισημάνατε κι εσείς. Το βασικό είναι να πλαισιώσουμε τη στρατηγική μας αποστολή με μια πτυχή και ασφάλειας ε, και, συγγνώμη, ασφάλειας και ανάπτυξης. Και νομίζω εκεί βρίσκεται η, η απάντηση. Στη χρηστή διακυβέρνηση, στην ε, δημιουργία των κρατικών δομών και των θεσμών υπάρχει μια πτυχή και εκπαίδευσης, γιατί αυτές οι χώρες έχουν μια ε, μεγάλη δημογραφική αύξηση Οπότε αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Γιατί αν δεν βρουν μέλλον στην πατρίδα τους θα στραφούν αλλού. Οπότε το G5 δεν ασχολείται μόνο με στρατιωτικά θέματα, με, αλλά και με στήριξη της κυβέρνησης, της κοινωνίας των πολιτών και επιστροφή του πληθυσμού. Επιστροφή του νόμου και της κυβέρνησης. Και ναι, μεν έχουμε πτυχές ασφάλειας και άμυνας, αλλά συστήσαμε και το καταπιστευματικό ταμείο που προσπαθεί να αντιμετωπίσει το θέμα της μετανάστευσης, διάσκεψη κορυφής βαλέτας, πολλά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν τα κράτη-μέλη. Και υπάρχει και το ενδυμικό πρόβλημα να φροντίσουμε να μην επαναλαμβάνονται τα προβλήματα που λύνουμε. Και στόχος είναι να διαπιστώσουμε κάποια στιγμή ότι σημειώθηκε πρόοδος και αυτή η πρόοδος να αξιοποιείται και να μην χάνεται. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ο κύριος Γκάλερ μίλησε για την ΕΚΟΒΑΣ, στις περιφερειακές δυνάμεις. Δηλαδή ρωτάτε γιατί οι Αφρικανοί δεν ασχολούνται με τα προβλήματά τους γιατί δεν προσπαθούν να ασχοληθούν οι ίδιοι με αυτά. Το επιδιώκουμε και θέλουμε να στηρίξουμε την δύναμη του G5, κάτι που είναι πρωτοφανέ, όπως το MGTF. Εκεί φαίνονται οι προσπάθειες των ίδιων των Αφρικανών. Και κάπως προκάλεσαν την Ηνωμένα Έθνη με τη σύσταση αυτής της δύναμης. Αποφάσισαν να δράσουν μόνοι τους και τώρα ζητούν βοήθεια. Αλλά και τα όρια της βοήθειας θα πρέπει να είναι οριθετημένα. Και επίση οι φιλοδοξίε να είναι λογικέ για να μπορούν να τύχουν και χρηματοδότηση και στήριξη. Και έτσι ο ρόλο των αφρικανικών περιφερειών στα πλαίσια του ΣΥΝΤΙΑ και του ΕΚΟΒΑΣ είναι κέριος. Το ΣΥΝΤΙΑ που είναι η περιοχή πιο ανεπτυγμένη με τα, τα προβλήματα στο Μαλί δεν έδρασε αποτελεσματικά παρόλα αυτά. Οπότε προσπαθούμε να ενισχύσουμε ε, τις περιφερειακές οργανώσεις. Αυτά ελπίζω να ήμουν αρκετά ακριβής, αλλά αν σας να απορίες, πολύ ευχαρίστω να συμπληρώσω. Σας ευχαριστώ. Και εγώ γιατί είναι τόσο ενδιαφέρουσα αυτή η ανταλλαγή απόψε. Ενημερώνω εσάς όσο και τους συναδέλφους ότι προς το τέλος του έτους θα έχουμε μια κοινή αποστολή μας με την ΑΦΕΤΑ για να επισκεφθούμε στην αιτήσα Μπέπα την ε, έδρα της Αφρικανικής Ένωσης και μετά θα πάμε και στον Ήγηρα. Αυτά. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερος για τη συζήτηση. Διάφορα. Ουχή. Σας ευχαριστώ και εύχομαι τις καλύτερες δυνατές διακοπές μετά το καλοκαίρι. Ξανασυναντιόμαστε. Ρώμηνα, Πολυκατάνια, Μεσόγειος είναι το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας. Καταγραφή ναυτικών προσπαθειών. Ευχαριστώ και γεια σας. to thank all interpreters, wishing you as well very best. Ευχαριστούμε πολύ και τους Γερμανείς, λέει ευγενικά η Πρόεδρος. Το αξίζει.